Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Welcome to the continuation of the AFET meeting. Καλημέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε με δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης που έχουν σχέση με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ξεκινώντας από το 24, ενημέρωση σχετικά με την αποστολή παρατηρητών στις εκλογές που έγινε στη Βοσνία Ζωγοβίνη στις 7 Οκτωβρίου. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι σε, στο πλαίσιο μιας διεθνούς αποστολής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ αποστήλαμε παρατηρητές στις εκλογές στη Βοσνία Ζωγοβίνη που έγιναν στις 7 Οκτωβρίου. Οι εκλογές αυτές είναι, ήταν πολύ σημαντικές για το μέλλον της χώρας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έγγελ, ότιμο μέλος της Επιτροπής μας, που ήταν επικεφαλής της ε, αποστολής των παρατηρητών. Μάρτιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Θεωρώ ότι μου κάνετε κοπλιμέντο. Λοιπόν, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Υποθέτω ότι διαβάσατε την έκθεση. Η Βοσνία, όπως ξέρουμε, δεν είναι η ευκολότερη χώρα στον κόσμο, δομικός. Να σας υπενθυμίσω το διακύβευμα των τελευταίων εκλογών είχαμε έξι εκλογές σε ένα. Αφορούσε την τριπλή προεδρία ταυτόχρονα, βουλευτικές εκλογές για την Ομοσπονδιακή Βουλή για την Ρεπούμπλικα Σέρψκα, την Βουλή της, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και για τα 10 καντόνια. Πολλές ε, κάλπες λοιπόν. Θα σας πω ε, ευθύ αμέσω πως αυτό το οποίο διαπιστώσαμε αλλά αυτά μπορεί να βρει κάποιος ε, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε παντού ήταν τα ίδια ευρήματα με τις αποστολές του ΟΑΣΕ και ήταν αρκετές αποστολές. Uh, uh, Κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γενικά λοιπόν και συνολικά καταλήξαμε ότι ήταν σχετικώς έφτακτες οι εκλογές και τυπικά ήταν σωστές. Μας είπαν όμως στις διάφορες ε, συναντήσεις ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Γιατί ο κόσμος από όλο το φάσμα της ε, κοινωνίας μας είπαν ότι υπήρξε ε, εντατική εκπαίδευση των ψηφοφόρων. Δηλαδή τους έλεγαν ε, το αμάξι σας, ε, το σπίτι σας, η δουλειά σας είναι ασφαλή μόνο αν κάνετε το σωστό. Αλλά αυτό συμβαίνει και αλλού. παρόλα αυτά, μια χώρα που έχει στόχο να γίνει υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ιδιωτός δεν θα είχε αυτά τα φαινόμενα μιλούσαν ε, για την ε, πιο βρώμικη προεκλογική εκστρατεία που είχε γίνει ποτέ και κατέστησε σαφές και σε εμάς ακόμα ότι οι περισσότεροι υποψήφοι δεν ε, ασχολούνταν με την Βοσνία Ριζεγοβίνη αλλά για την δική τους κοινότητα. Ε, αυτό φαίνεται ότι συνεχίζεται. Στο, παράγευο, στο Σαράγεβο πάλι σόκολατς ε, στην ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε ως μία μικρή αποστολή και θα ήταν ενδιαφέρον να πάμε πιο πολύ στην Ρεπούμπλικα Σέψκα γιατί την ίδια μέρα υπήρχαν μεγάλες ε, διαδηλώσεις ε, ανησυχούν των πολιτών για την εξαφάνιση και τον θάνατο δύο νεαρών που δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμα αλλά αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος και κατέβηκε στους δρόμους κατά δεκάδες χιλιάδες είναι ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί με το κράτος δικαίου. Αυτό το οποίο ακούγαμε είναι ότι οι άλλες χώρες έχουν τη μαφία και στην Βοσνία Ζεγοβίνη η μαφία έχει κράτος. Κάτι το οποίο μεταφέρει σχετικά ακριβώς την αίσθηση πολλών ανθρώπων που συναντήσαμε. Εντάξει, μπορούμε να λυπόμαστε τώρα, λυπόμαστε για διάφορα. Υπήρχαν διάφορες παρεμβάσεις στις εκλογές από γειτονικέ και όχι τόσο γειτονικέ χώρες. Αλλά βεβαίω η συμμετοχή συμμάχων από άλλες χώρες δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποκλείσουμε. Και βεβαίω ακούγεται κάπω περίεργο στους κατοίκου του Σεράγεβου να εμφανίζονται υψηλοί αξιωματούχοι της ε, Ρωσικής ομοσπονδία στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα. δεν ήταν χωρίς προβλήματα, αλλά σε γενικές γραμμές ε, ε, ήταν έφτακτη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι υπήρχε σοβαρή παρουσία εθνικών ε, παρατηρητών των εκλογών οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που είχαν κάνει μια συμμαχία για να παρατηρήσουν τις εκλογές υπό τον τίτλο Ποντλούπο και ήταν κάτι το οποίο βρήκα ενδιαφέρον. Υπήρχε μαζική προσέλευση χιλιάδων νέων που συμμετείχαν όχι ως υποψηφοί αλλά ως πολίτες για να παρατηρήσουν τις εκλογές. για να διασφαλίσουν την ορθή διεξαγωγή των εκλογών. Αυτά κύριε Πρόεδρε και βεβαίω οι λεπτομέρειες ε, είναι στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Τονίνο Πιτσούλα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Βλέπω ότι σας εκπλήσει αυτό. Δεν είχατε ζητήσει τον λόγο. Α, εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις εκλογές αυτές. Πρώτα απ' όλα, ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε επιτόπου αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, έχοντας ε, παρακολουθήσει εκλογές σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στην Αλβανία, στην Μακεδονία, στο Κωσυφοπέδιο. Ήταν σημαντικό να δούμε την κατάσταση και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη για να ολοκληρωθεί η παρατήρηση εκλογών σε αυτή τη λέσχη, ας το πούμε. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των παρατηρητών, σε γενικές γραμμές ήταν σωστές εκλογές. Παρότι δεν άλλαξε εντελώς ο πολιτικός νόμος. Ήθελα επίσης να πω ότι δεν εξεπλάγει από τα συμπεράσματα των παρατηρητών όσον αφορά ε, τον εθνοτικό κατακαιρματισμό και ε, την πόλωση. Ε, είδαμε ότι αυτή τη φορά η καταμέτρηση πήρε ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα και ότι η εκλογική περίοδος, η προεκλογική ξεκίνησε 1,5 χρόνο πριν. Είδαμε στη διάρκεια των συζητήσεων ότι υπήρχε αρνητική ρητορική, ε, ανέδει ο φόβος του παρελθόντος. Όλα αυτά δηλαδή ε, τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν ε, στο να μην υπάρχει αλλαγή και τα πολιτικά κόμματα να παραμείνουν ως έχουν. Βεβαίως υπήρχαν οι τιμένοι και υπήρχαν και οι κερδισμένοι γιατί έτσι τελειώνουν όλες οι εκλογικές διαδικασίες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συστάσεις και όταν θα έχει ολοκληρωθεί η έκθεση ε, της παρατήρησης των εκλογών ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς πάντα κάνουμε συστάσεις μετά από τέτοιου είδους παρατηρήσεις εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ε, Κοινοβούλιο και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Στην επόμενη επίσκεψή μου στο Σαράγεβο, που ευελπιστώ ότι θα γίνει αρχές Ιανουαρίου, ήδη θα αναφερθώ σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ράντοφ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da je dobro, da izvješća pokazuju da su izbori u tehničkom smislu Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που σύμφωνα με την έκθεση, έστω και από τεχνικής απόψεως, ήταν θετικές αυτές οι εκλογές αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν στην προεκλογική περίοδο. Δύο μπορώ να αναφέρω. Πρώτον, το σώμα, ε, το, το, η εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο και δεύτερο το θέμα της Ρεπούμπλικα Σέμπσκα. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα τριών ε, εθνοτήτων αλλά τελικά ε, έχουμε την περίπτωση όπου εκπρόσωποι ε, ενός τμήματος να εκλέγεται από άλλο τμήμα του πληθυσμού χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και κυρίως έλλειψη εμπιστοσύνης. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η Προεδρία ε, που θα πρέπει να έχει τρία μέλη εκπροσωπώντας τις τρεις εθνότητες. Ο Κροάτης εκπρόσωπος εξελέγει ε, από τα 2 ή 3% των ψήφων των Κροατών ε, πράγμα που δεν στέλνει καλό μήνυμα για τα δικαιώματα των Κροατών και πώς καλύπτονται αυτά στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, η Κεντρική ε, Εκλογική Επιτροπή ευελπιστούμε ότι θα προσπαθήσει να τα λύσει τα προβλήματα αυτά. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε τη Ρεπούμπλικα Σέρψη, έχουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη και έχουμε και την Ομοσπονδιακή οντότητα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν την δυνατότητα να λύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία έλαβαν χώρα και προέκυψαν πριν από τις εκλογές και το γεγονός βέβαια ότι και ο εκλογικός νόμος δεν άλλαξε. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να λυθούν για το μέλλον. Εδώ έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν είναι νόμιμη, δεν είναι νομιμοποιημένη υπάρχουν αποφάσεις του δικαστηρίου που λένε ότι ε, δεν έγιναν σεβαστές όλες οι αρχές κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ευχαριστώ κύριε Ράντος. Η κυρία Ζάφικο. Thank you, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά και η αλήθεια είναι ότι αναφέρομαι και μιλώ περισσότερο και στο κροατική συνιστό οντότητα της Βοσνίας Ρεσοκοβίνη. Πιστεύω, όπως και ο συνάδελφο έλεγε προηγουμένω ότι είναι πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο να αναδεικνύει όλα αυτά τα προβλήματα στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας έκανε προεκλογική εκστρατεία στην περιοχή ήδη ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Κροάτης ε, το συμπρόεδρος ε, έχει εκλεγεί με την υποστήριξη της Τουρκίας. Ε, έχουμε οδηγίες από θρησκευτικούς ηγέτες που λένε ότι ο Κροάτης συμπρόεδρος πρέπει να εκλεγεί από τους μουσουλμάνους. Κατά, κατά πλειοψηφία εξελέγει από τους μουσουλμάνους. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς όταν βλέπουμε την Τουρκία και τη Ρωσία να έρχονται στα σύνορά μα, στη σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για αυτέ τι εκλογέ σαν να είναι φυσιολογικέ. Δεν είναι φυσιολογικέ. Ε, πριν δύο μέρε, λίγε μέρε, είχαμε την ε, επέτειο των συμφωνιών του Ντέιτον. Ε, νομίζω ότι πρέπει σοβαρά να εξετάσουμε όλες αυτές τις επιρροές που προσπαθούν άλλα κράτη να επιβάλλουν στην περιοχή. Και ε, με εκπλήσει αρνητικά από όσο απόντες είμαστε ε, και πόσο δεν λαμβάνουμε στα σοβαρά αυτήν την περιοχή του κόσμου και την ε, ανάγκη να διασφαλίσουμε την ειρήνη σε αυτήν. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο πέραν από του κοινού συζητητέ. Όχι, από ό,τι βλέπω. Θέλετε, Μάρτιν, να ε, δευτερολογήσετε. Στην πρώτη μου παρέμβαση δεν μίλησα για θέματα περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, μιας και μιλούσαμε για παρατήρηση εκλογών, αλλά όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τις εκλογές πιστεύω ότι ξεχνάει το εξή, ότι ποιε είναι οι νομικέ δυνατότητε που υπάρχουν. Έγινε ό,τι έγινε, επειδή αυτό επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο της Βοσνίας Αρζεγοβίνης σήμερα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, έτσι ώστε το κράτος να λειτουργεί αποτελεσματικά και να είναι σύγχρονο. φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ίσω θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για να μεταβούμε σε ένα άλλο θεσμικό καθεστώ μετά τον Dayton. Ίσως να μπορεί να βοηθήσει προς αυτό και η Ευρωπαϊκή, Ένωση. Αλλά διαπιστώσαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της αποστολής ότι δεν υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στη χώρα αυτή για τη θεσμική της διάρθρωση από τους πολίτες για να έρθει αυτό πολύ και η Ιλιάνα. Ξέρετε, εάν έχουμε μία εκλογή στη Βαβαρία, το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό ο καγκελάριος της Αυστρίας να έρθει και να μιλήσει και να υποστηρίξει κάποιον υποψήφιο. Αυτό που μας ανησυχεί στη Βοσνία ριζογοβινη όμως, είναι ότι έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε την Τουρκία, έχουμε τους, ε, τη Σαουδική Αραβία, Και συνεχίζει να υπάρχει επίσης και μια λογική στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα που δεν επιθυμεί την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αν ποτέ η Βοσνία Ζεγοβίνη γίνει υποψήφια χώρα, θα χρειαζόμαστε να έχουμε έναν συνομιλητή, όχι δύο ή τρεις ή δυόμιση. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την ενότητα και το να έχουμε έναν συνομιλητή, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε υποψηφίου συμπροέδρου, ε, για παράδειγμα από την πλευρά των Σέρβων, οι οποίοι ανακοινώνουν πριν τι εκλογέ ότι αν εκλεγούν δεν θα έχουν διάθεση να συμμετέχουν στι ε, διαδικασίε. Φαίνεται ότι τελικά δεν θα το ακολουθήσει αυτό, αλλά έτσι έλεγε. Ε, εγώ ανησυχώ με την κατάσταση στα μίντια. Έχουμε, το έχουμε αναδείξει για το Κωσυφοπέδιο, για την Αλβανία. Δεν το έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε την Ισλαμική ουαπεχαμπιστική ε, επιρροή στη, στη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Όπως βλέπουμε πολλές ερωτήσεις παραμένουν ανοιχτές ακόμα. Θα μπορέσουμε ίσως να τις συζητήσουμε στο επόμενο θέμα τώρα, το οποίο αφορά την έκθεση, επί της έκθεσης της Κομισιόν για την Βοσνία Ζεγοβίνη για το 2018. Αυτή είναι η δεύτερη συζήτηση επί της έκθεσης αυτής. Καθώς η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να ζητήσω ε, από τον κύριο Πρέντα να μας παρουσιάσει τις κύριες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρέντα. Αυτή είναι η δεύτερη συζήτηση. Ξεκινήσαμε ήδη από τα τέλη Αυγούστου να συζητούμε ε, επί αυτής της νέας εκθέσεως. Ε, έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις από τότε ε, και μέσω των τροπολογιών που και εγώ ίδιος έχω υποβάλει προσπάθησαμε να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις εξελίξεις. Η τελευταία, το πιο σημαντικό μάλλον μεταξύ αυτών των εξελίξεων είναι οι εκλογές για τις οποίες μόλις συζητήσαμε. Επίσης συγκεκριμένες μάλλον θετικές εξελίξεις που θέλαμε να αναφέρουμε, όπως ας πούμε η έγκριση της στρατηγικής για την ενέργεια ή ακόμα και η πολλά αναμενόμενη τροποποίηση της ε, ε, νομοθεσίας. Ε, ε, εν ώψη των εκλογών. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες για θέματα τα οποία δεν μπόρεσα να, είχα, δεν μπόρεσα να αναφερθώ στην αρχική μου έκθεση γιατί είχαμε και κάποια προβλήματα με την μετάφραση. Ας πούμε, εξωτερική επιρροή για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ε, εκεί μια νέα παράγραφος όπου λέω ότι θα πρέπει να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη δέσμευση στην Βοσνία ε, για να επιτρέψει στη χώρα αυτή να προχωρήσει προς την ε, Ευρώπη και φυσικά να επιτύχει πολιτική σταθερότητα. 190 είναι οι τροπολογίες, δεν ξεπερνούν το μέσο όρο, είναι περίπου στο μέσο όρο. Δεν ε, έχει γίνει κάτι ρηξικέλευθο σε αυτή την περίπτωση. Και πρώτα Τινα και εγώ 27 συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν 124 τροπολογίες επί των 190 που έχουν υποβληθεί. Βεβαίω, προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερες απόψει, προσπαθώντας όμως να μην χάσω και την συνοχή της έκθεσης, γιατί καμιά φορά προσπαθούμε να βάλουμε όλα τα στοιχεία μέσα, ε, βάζουμε παραγράφους και ε, λέξεις και ε, φράσεις και μετά το σύνολο δεν. Είχαμε συνάντηση των Σκιωδών στο Στρασβούργο και τώρα ολοκληρώνουμε την εργασία επί των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστήσω τους ε, Σκιώδης εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν, αλλά και τον Τονίνο Πιτσούλα, ο οποίος ε, ήρθε ε, και δούλεψε μαζί μας ως επικεφαλής αντιπροσωπεία τη Επιτροπή που δουλεύει για την Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο. Δεν θα σας παρουσιάσω εν λεπτομερία τις 27 ε, συμβιβαστικές, όμως κάποια κεντρικά στοιχεία πρέπει να τα πω. Να πω εξ αρχής ότι είχαμε πολλές τροπολογίες για θέματα όπως είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα, η διακριτική μεταχείριση, η ελευθεροτυπία, η διαφθορά και η καταπολέμησή της, τρομοκρατία, εξτρεμισμός, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα σημεία αυτά επανέρχονται για μία ακόμα φορά και ε, βρίσκουν τη θέση τους στις, τροπο, στις ε, συμβιβαστικές. Επίσης εκτοπισμένοι και αγνοούμενοι μετά από την ε, σύγκρουση, μετανάστευση, θέματα πιο καυτά φέτος από ό,τι άλλες χρονιές το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος που επανέρχεται για μία ακόμα φορά. Τα κύρια μηνύματα τώρα των συμβιβαστικών Ευελπιστούμε ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη θα μπορέσει να σύμφωνα, ε, σύντομα συγγνώμη, να στείλει απαντήσεις στις ερωτήσεις που απευθύναμε έτσι ώστε να δούμε ε, ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε επί της υποψηφιότητας της χώρας. Δυστυχώς, δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαμε ακούσει στο Σαράγεβο. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουμε τις αρχικές απαντήσεις και το φθινόπωρο θα είχαμε απαντήσεις αρχές, αρχές Σεπτεμβρίου, μετά λίγο πιο πέρα, μετά λίγο μετά. Τώρα μας λένε ότι ενδεχομένως οι τρεις ε, πρόεδροι, ενδεχομένως λέω να έρθουν στις Βρυξέλλες, κομίζονται απαντήσεις. Θα το δούμε. Επανέρχομαι τώρα ξανά στις, ε, στους Ζητούμε λύση για την ε, ε, θέση σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των εκλογών. Τα είπαμε αυτά και λίγο πριν. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιτραπεί καμία προσπάθεια ε, μπλοκαρίσματος το, της συνταγματικής διαδικασίας. Επίσης, η τριμερής ε, προεδρία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης εγγενιάστηκε χθες. Από ό,τι κατάλαβα, το τέος μέλος ε, από την Κροατία ήταν στην Κροατία. Φαίνεται ότι ε, ε, πέρασε πολύ ωραία και γιορταστικά με τον πρέσβη της Ρωσίας και της Κίνας, άρα έχουμε κάποια κατεύθυνση εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όμως ακόμα πολλή δουλειά και πολλοί δρόμος παραμένει. Το μήνυμα το οποίο μπορούμε εμείς να στείλουμε σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον είναι το εξής ε, σε όλα τα επίπεδα ε, θα πρέπει οι αρχές να εκπαιδευτούν για να δουλεύουν υπέρ των πολιτών και για το συμφέρον των πολιτών όσον αφορά το δικαστήριο του λαού και της Ομοσπονδίας μετά από την υπόθεση Λούμπιτς ε, και ε, από το συνταγματικό δικαστήριο υπάρχει ένα νομοθετικό κενό. Σε γενικές γραμμές ε, υπάρχει πρόβλημα πολιτικής εκπροσώπησης στη χώρα. Ζητούμε λοιπόν εξέβρεση συμβιβασμών συμπεριλαμβανομένων και με την θέση σε εφαρμογή ε, των, ε, της απόφασης του δικαστηρίου για την υπόθεση Φίντσι και, και λοιπόν. Να σας πω το εξής. Έστω και αν εμείς ενστερνιστήκαμε την νέα προσέγγιση του 2014, ε, δεν σταματήσαμε ποτέ να ζητούμε την εφαρμογή της απόφασης αυτής και ζητούσαμε πολιτικές μεταρρυθμίσεις με την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμβιβασμού και συνένεσης. Και βεβαίως ε, οι συμβιβαστικέ μας τροπολογίες για μία ακόμα φορά αναφέρονται στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πολιτικές και κοινωνικές κλπ. Και αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για την ένταξη της χώρας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και σε κάποιες ιδέες, κάποιες πίστες έτσι ώστε ε, να δούμε πώς η χώρα μπορεί να το ευτιστεί με το ε, ακί, με το κεκτημένο. Αυτά εν συντομία ήθελα να σας πω. Οχτώ λεπτά, ε, δεν ήταν για το τέλος του κόσμου πια, λέει ο κύριος Πρέντα. Thank you very much. Now, next speaker is me. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπίτσουλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε αυτό το θέμα, να συντάξουμε αυτή την έκθεση που είναι απαιτητική. Κοιτώντα αυτό το προσχέδιο της έκθεσης για το 2018, πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν έτος εκλογών, επίσης ότι το συνταγματικό δικαστήριο χρειάστηκε να αλλάξει τον προεκλογικό κοινομοθεσία λίγο καιρό πριν τις εκλογές και επίσης ότι συνεχίζουν να υφίστανται τα χρόνια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη θεσμική αρχιτεκτονική αυτού του κράτους. Αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ε, έχουμε προσπαθήσει να εκπροσωπούνται όλες τις συνιστώσεις οντότητες, όλοι οι διαφορετικοί πληθυσμοί σε αυτή τη χώρα. Ε, ελπίσουμε ότι με το νέο εκλογικό νόμο θα επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα χρειαστεί από η Βοσνία Ερζεγοβίνη να μετασχηματιστεί σε ένα κράτος στο οποίο να σέβεται το κράτος δικαίου, στο οποίο να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση των πολιτών και Επίση θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα εκείνων των πολιτών που δεν ανήκουν σε κάποια από τις συνιστώσει ε, εθνότητες, όπως έδειξε η υπόθεση Φίτσι. Ε, οι συστάσεις των ε, εθνικών και διεθνών δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Ελπίζω ότι μετά τις εκλογές, θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό με τις νέες αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Εάν ε, συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κενό εξουσίας στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη, η κατάσταση θα γίνει χειρότερη. Θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια του 2018 δεν είχαμε πρόοδο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η κατάσταση παραμένει στάσιμη σε πολλούς τομείς και δυστυχώς ελπίζω η, με τη νέα Βουλή τη Βοσνία Ριζογοβίνης να έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε καλύτερα επί τη βάση της συμφωνίας σύνδεση. Είναι η μόνη ε, χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που ακόμα, για την οποία ακόμα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα τον, πρόεδρο, τον λόγο στον πρόεδρο της ομάδας εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, τον κύριο Κούκαν. Κυρίες και κύριοι, πέρασε άλλη μία πολλωμένη πολιτική εκστρατεία. Ελπίζω όμως η πολιτική ηγεσία να επιταχύνει την διαδικασία μεταρρυθμίσεων και την μεταρρυθμιστική ατζέντα ε, τα λέω, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα. Η έκθεση σημειώνει τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της οικονομίας αγοράς, ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της ελευθερίας έκφρασης. Η έκθεση αναφέρεται στις ε, παραβιάσεις των υποχρεώσεων της ε, συμφωνίας λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι της χώρας. Επιπλέον η χώρα δεν ε, εφαρμόζει τις αποφάσεις ε, του ΕΔΑΔ σε περιπτώσεις Βίσνατς, Πόλακ κτλ. Πρόκειται για σοβαρές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να αρχίσει να παίρνει σε σοβαρά η χώρα. Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά το να επενέσω εκείνα τα άτομα τα οποία προσπαθούν να ξεπεράσουν τους διχασμούς στην χώρα και δραστηριοποιούνται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα ήθελα να επενέσω τους μαθητές ε, του Λυκείου, του Βιάνιτσε, επειδή κέρδισαν το βραβείο Max van ε, ε, για τον ακτιβισμό τους. Διαμαρτυρίες στην Πάνια Λούκα για τον θάνατο του Ντραγκίτσεβιτς επίσης πρέπει να αναφερθούν. Πρέπει νομίζω να επενέσουμε αυτούς οι οποίοι παλεύουν για την ελευθερία έκφρασης ε, κατά α, της ρητορικής μίσους, ε, του θρησκευτικού μίσους ε, κτλ. Γι' αυτό νομίζω αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η Βοσνία Ζεγοβίνη, να γίνει μια σύγχρονη χώρα με έμφαση κυρίως στους πολίτες και όχι στις εθνοτικές ε, διαφορές. Ο κύριος Παπαδάκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη του αρκετές από τις τροπολογίες μας στους συμβιβασμούς και κυρίως για την έμφαση στην κοινωνική διάσταση που αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ορίζεται στη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι όντως σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία Ζεβοβίνη να προωθηθούν με ισορροπημένο τρόπο, με διαφάνεια και διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, με τρόπο ώστε να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των κατοίκων της χώρας, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας με την απαραίτητη προστασία για τους λιγότερο ευνοημένους στην κοινωνία. Αυτό είναι σημαντικό έτσι, έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να είναι μέτοχος σε όλη τη διαδικασία αλλά και οι νέοι να παραμείνουν στη χώρα και να πιστέψουν σε έναν ευγείονο μέλλον. Γι' αυτό τον λόγο ζήτησα χθε όπως υπάρξουν δύο μικρές αλλαγές στις συμβιβαστικές τροπολογίες 10 και 23 και πιο συγκεκριμένα την αλλαγή του λεκτικού στις τροπολογίες 98 και 172. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω, καθώς έχω αποστείλει σχετικό email στον κύριο Πρέτα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να αναδείξουμε και να τονίσουμε ακόμη περισσότερο ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας θα αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα θα επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί πολιτεύονται και θα δώσει ελπίδα για το καλύτερο μέλλον σε όλους τους πολίτες της χώρας ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση ή τη θρησκεία τους. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την πλήρη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι συνταγματικές και εκλογικέ μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμβαδίζουν. Οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας πολιτικής κουλτούρας βασισμένη στο συμβιβασμό και στην αμοιβαία κατανόηση. Κρίνεται αναγκαίο ότι οι κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσέγγισης με μεγαλύτερη όμως έμφαση στο European Pillar of Social Rights, όπως επίσης και η καταπολέμηση των στερεοτύπων στην κοινωνία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακόμη πιο σημαντικός αφού οφείλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Papadakis, Hvala lijepa gospodine Kukan. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Predi na e, dobroj suradnji. Sada e, se vhajstvo, ευχαριστήσω και τον κύριο Πρέντα για την εξαιρετική του έκθεση και συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι δεν θα πέρασε εύκολα μέχρι στιγμής. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο συνταγματικό ζήτημα. Ζητούνται συνταγματικές αλλαγές, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Χρειάζονται άλλοι μηχανισμοί πέρα από το να ζητάμε απλώς ε, αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Οι συνταγματικές αλλαγές ε, μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές ε, και στην συμφωνία του Ντέιτον, αλλά αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο πολιτικό ζήτημα. Η ε, εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων όσον αφορά την περίπτωση Σέιντι της Φίντσι, η αναγνώριση των συνταγματικών λαών, η περίπτωση Λιόμπιτσι, και η δυνατότητα να ψηφίζει ο κόσμος στο Μόσταρ και τα λοιπά. Πέρα από αυτές τις τρεις αποφάσεις υπάρχουν δεκάδες άλλες αποφάσεις ε, των δικαστηρίων που δεν εφαρμόζονται. Η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει τέσσερα παράλληλα δικαστικά συστήματα που δεν είναι εναρμονισμένα. Συχνά μάλιστα είναι αντιφατικά. Και πέρα από τις αδυναμίες ε, του δικαστικού συστήματος, αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν ένα αντιφατικό δικαστικό σύστημα, το οποίο απαιτεί περαιτέρω δράση από εμάς. Γιατί έτσι το σύστημα αυτό ε, γίνεται άπονομοποιείται ε, και δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών και έτσι αυξάνονται και εντάσεις στη χώρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικαστικό σύστημα για να υπάρξει μια αλλαγή στο μέλλον. Να προσπαθήσουμε να αναρμονίσουμε αυτά τα τέσσερα δικαστικά συστήματα και να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις ε, των δικαστηρίων. Και έτσι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία του κράτους συνολικά. Σας ευχαριστώ και ως Μπέγκε. Ο κύριος Μπέλτερ, ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα. Είχαμε καλή συζήτηση ως ε, σκιώδης εισηγητές. Ε, έχουμε μια κοινή προσέγγιση και διαβάζοντας την έκθεση αυτή μου θυμίζει τη δεκαετία του 90 όταν έκανα ανταποκρίσεις ως δημοσιογράφος και ήμουν αυτό της μάρτυρας του τρομακτικού πολέμου και των πολλών θυμάτων. και τις ε, συνομιλίες μου με τον κύριο Ντράκουλιτς, ο οποίος αρνήθηκε ότι ήταν άνθρωπος και μου έλεγε ότι είμαι μόνο Κροάτης. Και Αυτά, αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον τη Βοσνία τη Εγωμένη. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Now I give it floor to... Ευχαριστώ, κυρία Ζελένα Ζούφκα. Λέει η κυρία Ζόικο. Σας ευχαριστώ για τα ωραία οράματα που έχετε. Ε, εγώ ήμουν πρέσβης της Βοσνίας. επί σειρά ετών. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στη χώρα που αναζητεί την ψυχή της. Προσφάτως, ο Πρωθυπουργό της ε, χώρας μου αναφέρθηκε στο ζήτημα της Φωσνίας Ερζεγοβίνης και είπε ότι η συμφωνία του Ντέιτον ε, έχει παραβιαστεί και το πνεύμα της και ότι αναζητούμε μία λύση για την κρίση. Αυτό το συζήτησαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, την Δευτέρα που μας πέρασε και νομίζω ο Πρωθυπουργός μας, ο Αντρέ Πλέγκοβιτς, που ήταν και αυτός επικεφαλής αυτών των συναντήσεων, έχει αντιληφθεί ποιο είναι το βασικό πρόβλημα και οι αιτίες. Ίσως λόγω του εγωιστικού ζητήματος, επειδή έχουμε ε, μεγάλη κροατική κοινότητα. Υπάρχουν 500.000 πολίτες της Ένωσης στη Βοσνία ριζεγοβινη ε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στα σύνορα με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχουμε περάσει τέσσερα ψηφίσματα τα οποία είναι το μέσο μεταξύ δύο άκρων του να διασφαστεί η χώρα δηλαδή. Και βεβαίως ε, τα ψηφίσαμε όλοι στην Ολομέλεια και πρέπει να πιέσουμε την Κομισιό να τα εφαρμόσει. Αλλιώ δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να βρούμε νέα λύση. Ναι, να είμαστε ρεαλιστές. Οι ευρωπαϊκές λύσεις είναι ομοσπονδιακές ε, χώρες. Η μόνη ευρωπαϊκή λύση για τη Βοσνία Ζεκοβίνη είναι η ομοσπονδιοποίηση και ο σεβασμός των ψηφισμάτων μας και ο σεβασμός ε, των ε, συνταγματικών προβλέψεων και να γίνει σεβαστή η συμφωνία του Dayton μέχρι να αλλάξει. Σας ευχαριστώ, δεν ζητάει κάποιο άλλο τον λόγο, οπότε θα δώσω τον λόγο στην κυρία Μίκλα Ματουέλ, προϊστάμενο της ε, αρμόδιας ε, μονάδας στη Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα Καλωσορίζουμε την έκθεση Πρέντα, τα ευρήματα της οποίας συμπίπτουν με την έκθεση της Επιτροπής, αυτή που δημοσιοποιήσαμε τον Απρίλιο. Φαίνεται και από την έκθεση σας και από τη δική μας, ότι έχει διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσει η Βοσνία Ριζεγοβίνη, εάν θέλει να συνεχίσει στο δρόμο της προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη και έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα προετοιμάζουμε τη γνωμοδότησή μας για την αίτηση που έχει υποβάλει η Βοσνία Ερζεγοβίνη για ε, να ξεκινήσει η δικασία ένταξης. Που η γνωμοδότηση θα περιγράφει τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ανάμεσα στα οποία θα είναι τα θεσμικά και νομικά προβλήματα ε, και η θεσμική και νομική δομή της χώρας που δεν είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο. Μετά η πολιτική ηγεσία της χώρας θα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να λάβει μια απόφαση. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή που κάνει την επιλογή να κάνει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και αυτή τη στιγμή χρειάζονται κάποιες προσαρμογές προκειμένου η χώρα να γίνει συμβατή, το θεσμικό της πλαίσιο να γίνει συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία έχει κάνει την επιλογή να το πράξει αυτό. αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν στο δυνατόν γρηγορότερα, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη συζητούμε με την πολιτική ηγεσία της χώρας κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις και αργότερα βεβαίως θα συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα τις μεταρρυθμίσεις που θα περιγράφεται ότι χρειάζονται στην γνωμοδότηση της Επιτροπής. Όπως είπα, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να την βοηθήσει τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και να την υποστηρίξει για να βρεθούν λύσεις που να είναι συμβατές με το κοινοτικό κτημένο. Αυτό είναι ο ρόλος της Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια θα συνεργαστούμε και με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στα οποία φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να παίξει και θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εμείς ευχαριστούμε. είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ζητήσω τον κύριο Πρέντα να την συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν. Euh, euh, Όσον αφορά το ACPC, το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος Πίτσοβα, νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν μπλοκαριστεί για μία ακόμα φορά ε, η δημιουργία του CPC, ε τότε τι να πω. Το ανώτατο δικαστικό δηλαδή και εισαγγελικό συμβούλιο. Εγώ επέμεινα ε, όσον αφορά το θέμα αυτό ενώπιον όλων των υποψηφίων. Ακούω αυτά που λέτε κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τις εθνοτικές διαιρέσεις και το hate speech δυστυχώς δεν το έχουμε εκριζώσει και στις χώρες μας, κυρίως στις γειτονικές. Είναι γεγονός πάντως ότι στη Βοσνία Ζεγοβίνη αυτού του είδους το αφήγημα ε, μέσω μάλλον αυτού του αφηγήματος αναδύεται αυτόματα ε, και η μνήμη του πολέμου που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα να πω δύο λόγια σχετικά με αυτό που είπε η Ιρένα Ζόφκο. Τα μηνύματά μας δηλαδή. Νομίζω ότι τα μηνύματά μας ευθυγραμμίζονται με αυτά του Συμβουλίου και αναφέρθηκε άλλωστε ε, και η θέση του φίλου Πρέγκοβιτς στο Συμβούλιο τα μηνύματα είναι ίδια με τα μηνύματα του Συμβουλίου. Δηλαδή ότι θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να ε, ε, ε, τοποθετηθούν οι αρχές, να αρχίσουν να λειτουργούν, να αρχίσουν να υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις, αλλά βεβαίως πέρα από το τι λέμε εμείς, οι ίδιοι οι Βόσνοι θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν είμαστε εμείς διαπραγματευτές ΕΣΑΗ, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε προς όρασα. Αυτά σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και θα περιμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Thank you very much. That concludes the debate. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε μέσω παρατηρήσεων. Επόμενα θέματα. Τα επόμενα δύο σημεία αφορούν το Αφγανιστάν εξού και θα τα πάρουμε μαζί. Δηλαδή θα μας απασχολήσουν από κοινού θέλω να πω. E Έχουμε λοιπόν συμφωνία συνεργασία για την εταιρική σχέση για την ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν και ε, συμφωνία συνεργασία για την εταιρική σχέση και το, την ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Ε, το Αφγανιστάν εδώ και 40 περίπου χρόνια ε, αποτελεί πεδίο ε, ε, μαχών και αντιπαραθέσεων Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ε, την ε, ε, δέσμευσή της στη βελτίωση της κατάστασης και ως, ως προσεπίρωση μάλλον αυτών προχώρησε σε υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας για τη Δική Σκέψη. που τέθηκε σε ισχύ το 2017, ε, που όμως ε, δεν έχει ε, ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία ακύρωσης. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανοίξει δύο παράλληλες θέσεις. Πρώτον, ένα νομοθετικό ψήφισμα για τη διαδικασία, καθώς επίσης και άλλο ένα ακολουθών ψήφισμα για την συνολική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Φώτιγκα, αλλά δεν είναι εδώ. I see that Mr. Όμως ε, ο εκλεκτός συνάδελφος Ζαμπάσκι είναι εδώ και είναι ε, πρόθυμος να μιλήσει ε, στη θέση της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάω εξ ονόματος της συναδέλφου Φωτίγκα που είναι ε, αρμόδια για το θέμα αυτό και η οποία ζητά συγνώμη για την αδυναμία της λόγω ε, προβλημάτων υγείας να είναι σήμερα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μου ζήτησε να παρουσιάσω την γνωμοδότησή της. Πέμπτος χρόνος ε, μετατροπής, μεταρρύθμισης του Αφγανιστάν αυτή που ξεκίνησε το 2014 με την ε, απόσυρση των ε, διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων. Παραμένουν βέβαια πολλές προκλήσεις όσον αφορά την κοινωνία του Αφγανιστάν, ε, την ασφάλεια κλπ. Είναι σημαντικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Ε, χαμηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία, πολύ εκτοπισμένη λόγω των συγκρούσεων που δεν έχουν ακόμα σταματήσει. Η σύγκρουση ε, ε, εξεκολουθεί και με δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και ταλαιπωρεί ε, ε, σημαντικά ε, τον κόσμο, τους πολίτες που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τρομοκράτες και τρομοκρατικές ενέργειες. Εξού και είναι πολύ σημαντικό να είναι ενωμένοι οι ηγέτες έτσι ώστε να οδηγήσουν τη χώρα στην ασφάλεια και την σταθερότητα. Αυτό όμως θα καταστεί δυνατόν μόνον εφόσον σε μικρό επίπεδο, τοπικό επίπεδο αλλά και σε μάκρο ε, επίπεδο, ε, ακόμα και σε επίπεδο διεθνούς σκηνής, ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος του Αφγανιστάν, να βοηθήσει. Έτσι έχει λοιπόν η παρούσα κατάσταση στο Αφγανιστάν κάποιες ε, συστάσεις που θα μπορούσε να κάνει ε, για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ε, να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν, να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρτιση για την αντιτομοκρατία ε, και εκπαίδευση ε, σε ε, ίδιους τρόπους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Για τα οικονομικά τώρα. Η έκθεση αναφέρεται στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν τώρα. Επίσης διατυπώνει και δράσεις και συστάσεις τις οποίες μπορούμε να εμπλακούμε. Ας πούμε, υποστήριξη ε, των νέων ε, πολιτικών της κυβέρνησης, καταπολέμηση της ε, καλλιέργειας και προμήθειας ναρκωτικών κλπ να συνεχιστεί η κατάρτιση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των εγχώριων δυνάμεων. Δυστυχώς είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ε, αναφέρονται στην γνωμοδότηση και στα οποία θα πρέπει να δοθεί μία απάντηση. Μετά την ε, διάσκεψη στο Αφγανιστάν ε, ε, της 3ης Νοεμβρίου, καλό θα ήταν να τροποποιηθούν και τα σχετικά σημεία. Τέλος, η κυρία Φωτίγκα περιμένει και προσδοκά να συνεργαστεί με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και αναμένει εναγωνίως τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στους ομιλητέ. Πρώτος ο Αρνόντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάτι ήθελα να πω για την ε, γαλλική μετάφραση. Δεν είναι ο ΟΗΕ αυτός που εκπαιδεύει τις, ε, τα, τους, το στρατό του Αφγανιστάν, είναι το ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να το διευκρινίσω. Αυτό ναι. ήταν ένα λάθος στην γαλλική μετάφραση, λέει ο κύριος Θα είχα και πολλά να προσθέσω σε αυτή την έκθεση, όμως θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το ποια είναι η κατάσταση του Αφγανιστάν. Και αυτή δεν είναι καλή. Και από αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να ε, υπεκφεύγουμε. Στην ε, υποεπιτροπή τη οποία προεδρεύει η κυρία Φωτίγκα, είχαμε οργανώσει μια ακρόαση πριν λίγου μήνε και ακούσαμε τους εμπειρογνώμονε να μας εξηγούν ότι στην πραγματικότητα οι Ταλιμπάν δίνουν την εντύπωση ότι έχουν ισχύ, ε, αλλά στην πραγματικότητα είναι στα, στα, τελειώματα τους, δεν, δεν έχουν ε, και πολλές δυνατότητες ακόμα. Αλλά αυτό το ακούμε για χρόνια. Ε, δεν είναι η κατάσταση λοιπόν ελεγχόμενοι ε, στο πεδίο και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και να το τονίσουμε. Από την πλευρά των δικών μας προτεραιοτήτων. Βεβαίως πρέπει να προωθήσουμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση των ε, εμπορίων ναρκωτικών. Βεβαίως, ναι, αλλά αυτά τα λέμε από το 2001 ως προτεραιότητες για το Αφγανιστάν. Επομένως, βεβαίως και πρέπει να επαναβαβαιώσουμε την υποστήριξή μας στο στο, στη, στην πρόοδο που θέλουμε να δούμε για το Αφγανιστάν, αλλά πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και μια ρεαλιστική αίσθηση του τι μπορούμε να επιτύχουμε. Γιατί επίσης δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι συνομιλητές μας από το Αφγανιστάν έχουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση που θα χρειαζόταν για να πετύχουμε αυτά που λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με το εμπόριο των ναρκωτικών ιδιαίτερα και σε σχέση με τη διαφθορά ιδιαίτερα ορθά επισημαίνει η έκθεση παρόλο που το κάνει με πολλούς εφημισμούς και διπλωματικά, το ρόλο των όμορων χωρών. Είναι ένας ευγενικό τρόπος για να πει ότι οι γειτονικέ χώρες φαίνεται να μην επιθυμούν πάντοτε ένα ειρηνικό και ευημερούν Αφγανιστάν παίζουν ένα ρόλο αποσταθεροποίησης πολλές φορές ενεργά στο Αφγανιστάν οι χώρες αυτές. Και στην ενότητα στην οποία μιλούμε για την ε, τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία, η οποία είναι στα πρώτα της στάδια και πολύ εύθραυστη. Έχω δύο παρατήρησεις. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι δεν πρέπει να βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή τις, τους Ταλιμπάν μαζί με όλες τις υπόλοιπες ε, ομάδες τις τρομοκρατικές. Μιλούμε για τους Ταλιμπάν ως εξεγερθέντες και τους θεωρούμε συνομιλητές. Δεν είναι το ίδιο με μια τρομοκρατική ομάδα ε, την οποία για παράδειγμα δεν θα καλούσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επομένω, πρέπει πιστεύω να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στου Ταλιμπάν και άλλε τρομοκρατικέ ομάδε. Ε, το δεύτερο σε σχέση με την ερευνητική διαδικασία είναι ότι θα χρειαστούν ε, λέγεται ότι θα χρειαστούν ε, ξένες ειρηνευτικέ δυνάμεις για να επιβάλλουν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό θα είναι το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει η ίδια η ειρηνευτική διαδικασία. Επομένω θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς διατυπώνουμε αυτό το συμπέρασμα. Ε, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τα, κράτη, τα υπόλοιπα κράτη θα ήθελαν να συνεχίσουν να, να έχουν στρατό στην περιοχή όταν τα αποτελέσματα είναι τόσο άσχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Πιτσούλα για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ εκπροσωπώ τον κύριο Φρουντζουλίτσα. Ως ε, σκιώδης εισηγητής θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Φωτίκα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Πράγματι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλά ζητήματα όπως η μετανάστευση, η υγεία, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η τεχνολογία, καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, του ξεβλήματος χρήματος, ε, των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημαντικά σημεία. Υπάρχουν γύρω στα 10 εκατομμύρια άνθρωποι με ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και την ανάγκη για αποτελεσματική στήριξη από το κράτος για τα ζητήματα αυτά, με στόχο να διασφαλιστεί η παροχή υγεία σε ευπαθεί ομάδε, μεταξύ των οποίων οι γυναίκε, τα κορίτσια τα γυναικόπαιδα γενικώ. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί η αναπηρία και η πνευματική υγεία. Έχει μια αργή ανάπτυξη η χώρα το 2014 με την ε, απόσυρση των διεθνών στρατιωτικών ε, δυνάμεων, ε, όμως έχουμε μια επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης όπως αναφέρθηκε πριν, είναι μια καλή βάση για την περαιτέρω εργασία μας, αν και υπάρχουν κάποια μικρά σημεία που θεωρώ ότι πρέπει να έχουν περισσότερη ουσία. Όπως παράδειγμα το Σχάριν, κάποια ζητήματα που αφορούν τον αρνητικό ρόλο των γειτονικών χωρών στο Αφγανιστάν. Πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την αιρεσιμότητα και τον διάλογο με τους Ταλιμπάν να συνεχίσουμε να... τις προσπάθειες μας για να καταπολεμήσουμε την καλλιέργεια και το εμπόριο ναρκωτικών που τροφοδοτούν τους διάφορους ε, πολέμαρχους και κατσαπλιάδες στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αουστερβίτσιους για την Άλτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Φωτίγκα για την εξαιρετική της έκθεση, η οποία αποτελεί μια καλή βάση για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις μας και θεωρώ ότι η περαιτέρω συνεργασία στον αναπτυξιακό τομέα καθώς υπάρχει και ένα δεσμευτικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντική για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Αφγανιστάν και αυτό φαίνεται και στο κείμενο που παρουσίασε η κυρία Φωτίγκα. Μάλιστα, Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτά σχετίζονται και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου πέρσι και συμφωνώ με τις εκτιμήσεις του συναδέλφου Ντανζόν για την ειρνευτική διαδικασία και την επίτευξη μιας ε, σταθεροποίησης στο Αφγανιστάν. Οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί να βρούμε διάφορους εταίρους ε, και γείτονες. Αλλά και πάλι η ειρήνη είναι η μόνη απτή λύση για μια σταθεροποίηση της χώρας. Ε, πρέπει να εμπλακούμε γνωρίζοντας ότι θα είναι δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους μας και την Ειρηνευτική Συμφωνία. Έχοντας αυτά κατά νου, συνάδελφοι, θα πρότεινα να εμπλουτίσουμε την έκθεση της κυρίας Φωτίγκα με κάποιες τροπολογίες. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη έμφαση στο πλέγμα ασφαλείας και τα προαπαιτούμενα ε, για να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας, ανάπτυξης, ε, φτώχειας, ε, ανάπτυξη πέθρου, ανθρώπινης ανάπτυξης, κατά προτεραιότητα. Δεύτερον, η περιφερειακή διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα πρότεινα κάποιες τροπολογίες που αφορούν την περιφερειακή διασύνδεση. Κάποιες χώρες Κεντρικής Ασίας έχουν μεγάλα έργα, όπως ξέρετε, για να κατασκευάσουν τεράστια έργα υποδομών. Και αυτό το σημαντικό στοιχείο νομίζω θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο κείμενο. Όταν μιλάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια δεδομένων των πόρων που στέλνουμε στο Αφγανιστάν. Να σας πενθυμίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής με 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς να μετράμε τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, θα πρότεινα να υπάρχει μια πιο αναλυτική αξιολόγηση των βουλευτικών εκλογών που όπως ξέρουμε έλαβαν χώρα στις 27 ε, Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευτεί και δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Αλλά πρέπει νομίζω να αντικατοπτρίζονται. Και θα καλύψουν επίσης οι τροπολογίες μου το θέμα της ε, αυξανόμενης βίας των ε, Ταλιμπάν τους βιασμούς, τα δικαιώματα των γυναικών, τα ναρκωτικά και τους ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους. Που θα πρέπει να εξοριχθούν με τρόπο διαφανή. Και αναμένω τη συνεργασία με την Αναφωτήγκα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βαλέρο για τους πράσινους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση της κυρίας Φωτίγκα. Ε, ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ότι η κατάσταση είναι εσχίστη ε, στο Αφγανιστάν και δεν βελτιώνεται. Αυτό πρέπει να αναφερθεί ξεκάθαρα στην ε, έκθεση. έστω και εάν ε, γίνεται κάποια αναφορά ε, ε, ακροθυγός στο θέμα της κοινής, του κοινού θέματος των μεταναστών, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα της μετανάστευσης που προέρχεται από τη χώρα αυτή, ενώ εδώ δεν γίνεται ιδιαίτερος λόγος γι' αυτό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης του Αφγανιστάν μίλησε στην Σουηδική τηλεόραση και ζήτησε να μην επιστρέφονται στη χώρα ε, ε, οι νέοι Αφγανοί διότι δεν είναι ασφαλής η χώρα. Η Σουηδία ε, φαίνεται να είναι η χώρα που έχει επιστρέψει ε, ε, τις περισσότερες, τους περισσότερους νέους στο Αφγανιστάν. 53 παιδιά πρόσφατα από τη Γερμανία, από την Νορβηγία και από την Σουηδία έχουν σταλεί πίσω στην χώρα τους, στο Αφγανιστάν. Αλλά αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από τους Ταλιμπάν ή από εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα αυτή. Εμείς βεβαίως ξεκινήσαμε να υποβάλουμε προσφυγές ε, για το θέμα αυτό. Αλλά, αλλά ε, θα πρέπει ε, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Το Αφγανιστάν, να μην ξεχνάμε ότι ε, υποδέχεται και μετανάστες ε, από χώρες γειτονικές. Και το Αφγανιστάν επανειλημμένα έχει πει ότι δεν αντέχει να ε, περιθάλψει όλους αυτούς τους ε, ε, πρόσφυγες. Ε, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν γιατί πραγματικά το, ξανα, το είπε και ο υπουργό και το έχουν πει επανειλημμένα ότι δεν τα καταφέρνουν να, να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των προσφύγων. Βεβαίως ε, μερικοί πιστεύουν ότι το, και ένα άλλο πρόβλημα θέλω να, να ε, αναφέρω, ότι ε, στην διεθνή σκηνή είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι το Αφγανιστάν είναι μια ενιαία χώρα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι πολλές οι εθνικές ομάδες, ομάδε, ομάδες, οι οποίες αντιτίθενται η μία στην άλλη, διαφορετικές ομάδες, οι των και άλλων που με μετακινούνται μάλιστα και εντός της χώρας πρέπει να ε, αποφύγουμε, ε, ας πούμε οι Άζαροι μεταξύ των μουσουλμάνων, να φύγουν από το Αφγανιστάν. Επομένως, το μέλημά μας όσον αφορά το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να είναι μονάχα στρατιωτικό, αλλά θα πρέπει να είναι και κοινωνικό, θα πρέπει να είναι και πολιτιακό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία, γιατί διαφορετικά θα πέσουν στα νύχια των Ταλιμπάν, θα πέσουν στα νύχια των εγκληματικών οργανώσεων. Εν σε περιπτώσει εγώ θα υποβάλω τροπολογίες, γιατί θεωρώ ότι η έκθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει και τα στοιχεία αυτά. Thank you very much. Next speaker. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λέζι, μέρος της ΓΚΟΕ. Ε, ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Είναι θετικό ότι μιλάμε για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών, την ισότητα των φύλων. για έναν διάλογο και συνεργασία βεβαίως Βεβαίω, ε, όπως είπε και ο κύριος Νταζάν, υπάρχει ο κίνδυνος ε, οι στόχοι αυτοί να είναι διφορούμενοι. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά σε κάποιο ορατό μέλλον. Αλλά το ερώτημά μου είναι εάν ε, η κατεύθυνση των μέτρων αυτών που παρουσιάζονται στην έκθεση ε, θα μπορούσε να είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να επιτευχθούν κάποτε αυτοί οι στόχοι. Παραδείγματος χάρη ε, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με αυτόν του δημοσίου τομέα. Παραδείγματος χάρη στο άρθρο 18 για ε, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και δημοπρατήσεις ε, εκεί πέρα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι φορείς του ιδιωτικού τομέα. Και εκεί και στο άρθρο 37 για τους φυσικούς πόρους, ειδικά στον εξορυκτικό τομέα, να υπάρχει διαφάνεια στις άμεσες ξένες επενδύσεις, να δημιουργηθεί ένα απαραίτητο πλαίσιο. Επίσης, ε, τα ζητήματα εμπορίου των φυσικών πόρων. Αυτά είναι μέτρα συνεργασίας με άλλες ε, χώρες, ε, στα οποία έχουμε μεγάλες εμπειρίες, οι οποίες δεν είναι πάντα θετικές. Και δεν ευνοούν πάντα τη βελτίωση της κατάστασης για όλο τον λαό. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Ε, αυτό ακριβώς θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξουν προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Οι φυσικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, ώστε να ωφελείται πρώτα απ' όλα ο αφγανικός πληθυσμός. Και ε, πράγματι εξηγήθηκε η κατάσταση, είναι καταστροφική. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ είναι περισσότερο μέρος του προβλήματος ε, παρά της λύσης. Και δεν συνεισφέρει στην ειρήνη και την ασφάλεια. και όπως ε, και η κυρία Βαλέρο, έτσι και εγώ ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Στο θέμα του άρθρου 28 αναφέρθηκε η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης. Εδώ πέρα θα ήθελα μόνο να πω ότι αυτό έχει ως στόχο τη σύναψη μιας συμφωνίας επανεισδοχής. Τα είπε η κυρία Βαλέρο. Είναι ανεύθυνο νομίζω να στέλνουμε πίσω σε αυτή τη χώρα ανθρώπους. και θα ήθελα να το τονίσω, δεν θα πρέπει να δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια με όρους για το μεταναστευτικό. Και θα καταθέσουμε τροπολογίες ε, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλιομάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω ότι ο συνάδελφος ε, πρέπει να τη συγχαρούμε για το εξαιρετικά ισορροπημένο κείμενο που μας παρουσιάζει. Έχω λίγες παρατηρήσεις. Παρά το γεγονό ότι πολλά είναι τα αρνητικά στοιχεία, πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και ένα θετικό, ότι υπάρχει συμμετοχή στι εκλογέ και θα πρέπει ιδιαίτερα να πούμε ότι ε, και για να είναι κανεί υποψήφιο και για να συμμετάχει στι εκλογέ πρέπει να είναι πολύ θαραλέο στο Αφγανιστάν. Επομένω πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Μετά, συνεχίζοντα τη σκέψη του συναδέλφου Αχνονταζόν, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ανάμεσα σε αυτά προβλήματα με τα οποία δεν αναδεικνύουμε, όπως για παράδειγμα η σχέση μεταξύ των εθνοτήτων στο Αφγανιστάν και επίσης η παρέμβαση του Πακιστάν σε αυτές τις ε, συγκρούσεις ε, στο Αφγανιστάν, η οποία έχει ε, επιπτώσεις σε διάφορες περιοχές θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Αφγανιστάν παραμένει η καταπολέμηση του εμπορίου των ναρκωτικών. Αυτό, ε, το οποίο τελικά αυτό το, το εμπόριο των ναρκωτικών είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομία του Αφγανιστάν. Και στην καταπολέμηση του εμπορίου των ναρκωτικών μέχρι στιγμής έχουμε μόνο διακηρύξεις. Πρέπει να δούμε αποτελέσματα χειροπιαστά. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και μέτρα τα οποία θα αντικαταστήσουν την οικονομική σημασία που έχουν τα ναρκωτικά. Πρέπει να δώσουμε άλλε εναλλακτικέ στον κόσμο. Ε, αν δεν συμβεί αυτό δεν θα σταματήσει το εμπόριο των ναρκωτικών. Και επίση είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο τη κυβέρνηση για να αντιληφθούμε πώ λειτουργούν τα πράγματα στο Αφγανιστάν. Αυτό έχει επιπτώσει και στο πολιτικό επίπεδο, το οποίο σημαίνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύσει τη βοήθειά της με βάση αυτά που γνωρίζει για τη διαφθορά και για την κατάσταση επιτόπου και να στοχεύσει τις δράσεις της προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Επί χρόνια δίνουμε χρήματα ε, για μεγάλες υποδομές σε εθνικό επίπεδο, αλλά αν πάτε σε ένα χωριό, και εγώ έχω επισκεφθεί πολλές φορές χωριά στο Αφγανιστάν, αυτό που θα ακούσετε είναι γιατί να χρειάζεται να κάνουμε κάθε πρωί ε, μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων για να βρούμε νερό. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα εκεί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, πηγές ε, για το νερό, αλλά σε αυτές δεν έχουν πρόσβαση οι γυναίκες. Ή μπορεί να υπάρχει ιατρική περίθελψη από προγράμματα των, των, των γιατρών του κόσμου, αλλά αυτά να είναι πολύ απομακρυσμένα. Χρειάζεται λοιπόν συγκεκριμένε δράσει που να βοηθούν τον τοπικό πληθυσμό. Και τέλο, όσον αφορά τη στρατιωτική παρουσία, θα έλεγα ότι όλο και λιγότερε είναι οι χώρε που να επιθυμούν να στείλουν στρατό στο Αφγανιστάν. Εξάλλου, όταν παραμείνει μια στρατιωτική δύναμη πολύ ε, καιρό σε μια περιοχή, αρχίζει να εμφανίζεται σαν δύναμη κατοχής και να δημιουργούνται προβλήματα με τη σχέση της με τον τοπικό πληθυσμό. Ε, κάνουμε προγράμματα εκπαίδευσης του στρατού του Αφγανιστάν, αλλά αυτά δεν επαρκούν, δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί αυτοί οι οποίοι περνούν την εκπαίδευση τη στρατιωτική, μετά στρατολογούνται είτε από τους Ταλιμπάν, είτε από τους πολέμαρχους, είτε από άλλε τρομοκρατικέ ομάδε ή χρησιμοποιούνται στο εμπόριο των ναρκωτικών. Και αυτό είναι ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι διακηρύξει που κάνουμε δεν αρκούν. Ε, για να λύσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα του Αφγανιστάν θα πρέπει να κάνουμε χειροπιαστέ ενέργειες οι οποίε να απευθύνονται στην πραγματικότητα στο, στο πεδίο του, του πληθυσμού στο επιτόπου. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει εκπρόσωπο τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Εάν πράγματι ισχύει αυτό, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξωτερικών για το σχέδιο έκθεσης. για την σύμφωνη γνώμη στην Συμφωνία Συνεργασίας με το Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μακροχρόνια δέσμευση προς την χώρα και τον λαό της και θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ένας αξιόπιστος εταίρος έχοντας ε, βεβαίως ε, κατά νου το εξής ε, Υιοθετήσαμε και την στρατηγική για το Αφγανιστάν και πριν από μία εβδομάδα το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα του Συμβουλίου όπου εκφράσαμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Η Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική συμφωνία, είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε η στρατηγική μας να περάσει το επόμενο βήμα. Και μέσω της ε, προσωρινής εφαρμογής υπάρχει ήδη διάλογος για πολλά ζητήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση της έκθεσης ε, και κάποιες από τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα. Πράγματι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, αλλά από την πλευρά την δική μας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την προώθηση της ε, ειρήνης και την σταθερότητα στην χώρα αλλά θα εργαστούμε και για μια περιφερειακή συνένεση για την ειρήνη, η οποία, όπως τονίστηκε, έχει κέρια σημασία για να υπάρξει ειρήνη. Απέχουμε τώρα μία εβδομάδα από την αποστολή στην Γενέβη και θα υπάρξει ένας απολογισμός ε, των όσων συνέβησαν από την τελευταία μας συνάντηση πριν από δύο χρόνια. Και στην Γενέβη θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και με διεθνείς εταίρου για να προωθήσουμε την ειρήνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις ε, δράσεις μα και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να παραμείνει συνδεδεμένο και να παρακολουθεί το διάλογο αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, εισηγητή αν θέλει να πει δύο λόγια και να συνοψίσει την συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Είναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της κυρίας Φωτίγκα για όλες τις ε, ε παρατηρήσεις. Ε, οπωσδήποτε ε, θα, θα τις γνωστοποιηθούν, θα τις μεταφέρω ε, και είμαι βέβαιος ότι θα τις λάβει υπόψη της. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τη συζήτηση για αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη και τώρα... Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυργιζίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, υπαριθμών 28, ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών ε, της Κυργιζίας, κύριο Μπεκόφ Κυργίζ Αζαρματόβιτς. Κύριε Υπουργέ, Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να πω ότι η Κυργιζία είναι μία από τις αναδυόμενες δημοκρατικές χώρες της περιοχής. Βεβαίως ε, όλα δεν είναι, ε, ε, όλα δεν είναι θετικά, ωστόσο οι, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση βαθαίνουν όλο και περισσότερο. Πρόκειται για μια ε, ε, χώρα για την οποία ε, είναι έτοιμη μία πρόταση χρηματοδότησης από το 2021 και μετά που είναι πολύ σημαντική ταυτόχρονα διευρύνει την συνεργασία της η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την περιοχή μέσω ε, νέων μορφών συνεργασίας και εργαλείων συνεργασίας με τη χώρα σας. Η Επιτροπή μας προετοιμάζει σύσταση για το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς επίσης και την ύπατη εκπρόσωπο όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε τη σχέση καθώς επίσης και την πρόοδο που θέλουμε η σχέση αυτή να έχει έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να επικυρώσει τη συμφωνία όταν θα έχει ολοκληρωθεί. Κύριε Υπουργέ, σας δίνω τώρα το λόγο έτσι ώστε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Ξέτοιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στην Κυργυζία και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά μια νέα μορφή συνεργασίας. Ε, η κυριαζική πλευρά αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την συνεργασία που θεωρούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θεωρούμε σημαντικό εταίρο. Επίσης, συμφωνούμε με τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Ε, αξιολογούμε θετικά την ε, διαρκή ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δημοκρατία της Κυργιζίας, η οποία από την πλευρά της είναι δεσμευμένη για αποτελέσματα. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν, υπάρχει διάλογος μέσω συγκεκριμένων υποστηρικτικών εργαλείων τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δείξει την δέσμευσή μας ε, για ε, καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε ε, διότι ο κύριος Σόρο Τζιμπίκοφ, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κυργιζίας, τον Απρίλιο θα είναι εδώ ε, έτσι ώστε να ε, γίνουν διαπραγματεύσεις ε, και με τον κύριο Ταγιάννη και με άλλους επικεφαλείς θεσμικών οργάνων με θέματα διμερούς συνεργασίας. Επίσης, χαιρόμαστε γιατί η κυρία Μογκερίνη είπα ότι εκπρόσωπο τον Νοέμβριο του 2017 επισκεπτόμενη τη Δημοκρατία της Κυργυζία, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, ε βουλευτές, ε, η Δημοκρατία της Κυργυζία οδεύει στον δρόμο της δημοκρατίας ε, και του κράτους δικαίου μέσω δε των διαφανών γενικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2016 εγγράφηκε στην πορεία αυτή ότι Επίσης, έγιναν, έγινε δεκτή η νομοθέτηση αλλαγών στο συνταγματικό ε, στο, το, στο σύνταγμα της ε, χώρας σε σχέση ε, με τον τρόπο διακυβέρνησης και η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας από τον ένα πρόεδρο στον άλλον ε, σηματοδότησε την δημοκρατική εναλλαγή. Τα αποτελέσματα των εκλογών έγιναν δεκτά και από τη χώρα και από την διεθνή κοινότητα. Πρόσφατα εγκρίναμε ε, και στρατηγική ανάπτυξης ε, για τα έτη 14-18.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 ε, ολοκληρώσαμε μάλλον τη στρατηγική 14-18 ε, ε, για την ανάπτυξη της χώρας που περιλαμβάνει στοιχεία ανάπτυξης οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και επίσης αναφέρεται και σε ενδιάμεσα βήματα μια συνολικής στρατηγικής, ενός συνολικού στρατηγικού οράματος. Αγαπητοί βουλευτές, εδώ και 20 χρόνια η αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Κυργιζίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση των διμερών μας ε, σχέσεων ε, και οι προτιμησιακές ε, σχέσεις και η πρόσβαση και ένταξη της Κυριγιζίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σχέσεις όσον αφορά εσωτερικά θέματα και όπως η δικαιοσύνη, η πολιτισμός κλπ. αλλά και εξωτερικά θέματα ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικά. Ε, ε, ε, αξιολογούμε θετικά και εκτιμούμε την προσπάθειά σας όσον αφορά την νέα τη νέα εντολή για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κυργιζίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο είχε την εξέβρεση λύσεων αμοιβαίως ικανοποιητικών για τις δύο πλευρές. Ε, στην ε, διάρκεια της ε, επίσκεψης του Προέδρου τον Απρίλιο του 18 ε, στις ε, Βρυξέλλες ε, ξεκίνησαν οι βάσεις για μια ενισχυμένη συνεργασία και ένα νέο σύμφωνο συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα διεθνή κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές τάσεις, το σύμφωνο συνεργασίας αναφέρεται στην δημοκρατία της με τρόπο ε, ιδιαίτερα, ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Τον Δεκέμβριο ε, του 2017 ε, στις Βρυξέλλες είχαν μια πολύ καλή συνεργασία και ολοκληρώθηκε μέχρι τώρα ο πέμπτος ε, ε, γύρος. Το 18 τρεις ε, θεματικές ομάδες δουλεύουν με πολύ δραστηριο τρόπο και έχουν επιτύχει πολλά αποτελέσματα. Στην πρώτη θεματική συνεργασία οι αντιπροσωπείες επιτυχώς ολοκλήρωσαν εργασίες που κάλυψαν το 19% του κειμένου. Ταυτόχρονα υπήρξαν προβλέψεις ε, σχετικά ε, ε, με σημαντικούς οργανισμούς της Δημοκρατίας της Κυργιζίας και που παραπέμπουν στην ε, διεθνή διάσκεψη για το ε, δίκαιο, το ε, ποινικό δικαστήριο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής Συνεργασίας. Όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η Δημοκρατία της Κυργιζίας τον έχει υπογραφεί η συμφωνία αλλά δεν έχει επικυρωθεί και δεν εφαρμόζονται λοιπόν όλα τα στοιχεία ε, και δεν εφαρμόζονται λοιπόν όλα τα στοιχεία του καταστατικού της ε, Ρώμης ε, για την δημοκρατία της Κυργιζίας. και επομένως δεν ισχύουν και όλες οι διατάξεις οι οποίες στο καταστατικό αναφέρονται. Ε, ωστόσο υπάρχει ανάγκη για ε, ενδελεχή ανάλυση όλων των ε, στοιχείων έτσι ώστε να δούμε αν και κατά πόσο συνάδουν με την εσωτερική ε, νομοθεσία. Όσον αφορά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο συμμετείχε η Δημοκρατία της Κυργιζίας στην διάσκεψη και αυτή τη στιγμή τελειοποιείται από εμπειρογνώμονες ε, η θέση μας ε, ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Επίσης, τα αρμόδια σώματα θα συζητήσουν το θέμα όσον αφορά την επόμενη θεματική διαπραγμάτευση και συνεργασία. Υπήρξαν συνεφωνίες όσον αφορά το 90% του κειμένου. Ένα από τα αντιφατικότερα σημεία είναι το θέμα της ε, σύγκλησης ε, και της εναρμόνισης ε, της εθνικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κυργιζίας με την ενωσιακή νομοθεσία. Για την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρείται ως βάση των σχέσεων για, τα, για τους διάφορους οργανισμούς. Ωστόσο υπάρχουν κεφάλαια όπως ο συντονισμός, η πληροφόρηση των καταναλωτών, η προστασία των καταναλωτών, διασυνοριακή συνεργασία, επικοινωνία κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν. Όσον αφορά την δεύτερη θεματική ε, ομάδα, ε, για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα, πολλά ζητήματα παραμένουν ακόμα ασυντόνιστα ε, βάσει της ε, αρχικής ε, θέσης κάποιων οργανισμών της Δημοκρατίας της Κυργιζίας. Υπάρχουν ακόμα πολλά κεφάλαια όπως είναι η διανοητική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, τεχνικά προσκόμματα στο εμπόριο, επίλυση διαφορών, επενδύσεις κλπ. Αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανασυζητηθούν περαιτέρω. Η Δημοκρατία της ε, με ε, έχει καλύψει τις ε, υποχρεώσεις της με αφοσίωση όσον αφορά τις περιφερειακές, τους περιφερειακούς οργανισμούς. Ε, αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά ε, την, το σχέδιο συμφωνίας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εσωτερικές αρχές της EAU. Ιδιαίτερα συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τρία σημεία. duties, section of Κατασκευθέντα αγαθά όσον αφορά το εμπόριο, αυτό είναι ένα θέμα της Ευρασιατικής Οικονομικής ε, Επιτροπής. Ε, ε, κύριες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία σε επίπεδο επί κοινοβουλίων με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, υπάρχει και η ε, Επιτροπή για την Μογγολία και την ευρύτερη περιοχή και μας ενδιαφέρει η συνέχιση των συζητήσεων και η ανταλλαγή εμπειριών και βελτίστων πρακτικών. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της διεπιστήμης της ε, διακοινοβουλευτικής ε, συνεργασίας ε, μπορεί να προωθηθεί και το περιεχόμενο των κειμένων της, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς το 2014 γίναμε δημοκρατικός εταίρος, περάσαμε σε αυτό δηλαδή το επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ε, και την εμπειρία και το παρελθόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στις, και στο εσωτερικό μας. Η Κυργιζία είναι μία από τις μοναδικές χώρες της περιοχής με λειτουργών κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας αξίζουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαιτέρως ε, αξιολογούμε την τεχνική και λοιπή υποστήριξη προς τη δημοκρατία μας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το πολιετές ενδεικτικό πρόγραμμα ε, για την περίοδο 14-20 καθώς επίσης και το ενδεικτικό ε, πρόγραμμα για την Κεντρική Ασία ε, για την αντίστοιχη περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, θα πρέπει ιδιαίτερως να χρηματοδοτηθούν και να υποστηριχθούν προσπάθειες για το κράτος δικαίου κλπ. Ήδη σημαντικά επιτεύγματα έχουμε και αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο να συνεχίσει η υποστήριξη των ε, ε, θεμάτων όπως είναι ε, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος και του συστήματος των οργανισμών ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης προγράμματα όπως η παροχή πόσιμου ύδατος σε αγροτικές περιοχές, περιοχές της υπαίθρου να συνεχιστούν. Επίσης, ο κύριος Σόλον το 2018 ε, αναγόρισε το έτος 18 όσο το έτος της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου για την ε, χώρα μας. Αναμένουμε λοιπόν ε, περαιτέρω να, ε, στη διάρκεια του έτους και του επόμενου έτους ε, να προχωρήσει το Σύμφωνο Συνεργασίας Εταιρική σχέση και Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτεραιότητες θα πρέπει βέβαια και για το εξειδικευμένο στοχευμένο πρόγραμμα του επόμενου έτους να ε, αναφέρεται σε το πρόγραμμα που έχει ήδη οργανωθεί για το 18 με 20. Υπάρχει ήδη το Συμβούλιο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προεδρεύω εγώ και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την παρακολούθηση των έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυργυζή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η χώρα μας καλωσορίζει την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία που θα εγκριθεί του χρόνου χαιρόμαστε για το ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε ένα συνεχής και επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των χωρών της περιοχής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βασικούς τομείς αυτής της στρατηγικής, όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, εκπαίδευση, περιβάλλον και υδάτινη πόρη. Η χώρα μας ε, στηρίζει την ε, πλατφόρμα συνεργασίας με την Κεντρική Ασία. Αύριο 23 ε, Νοεμβρίου θα έχουμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ε, των δύο περιοχών υπό την ηγεσία της κυρίας Μογκερίνη. Επίσης, η Κυργυζία συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Ο ε, τελευταίος γύρος αυτού του διαλόγου ήταν στις 8 Ιουλίου στο Αζαμπάτ. Ε, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξή της όσον αφορά θέμα το οποίο έχει προκύψει από την εξόρυξη ουρανίου στην Κεντρική Ασία. Είχε οργανωθεί μια διάσκεψη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον. Στις 8 Νοεμβρίου φέτος ε, η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών για το θέμα αυτό οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΠΕ στο Λονδίνο, την ΕΤΕΠ. Οργανώθηκε και εκεί πέρα ακριβώς ε, το πώς θα μπορέσουμε να αφιερώσουμε οικονομικούς πόρους ε, για την βελτίωση του περιβάλλοντος της Κεντρικής ε, Ασίας. Ακριβώς για να λυθεί το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει από την εξόριξη ουρανίου. Προτείνουμε να εγκριθεί ένα νέο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας για να προληφθεί η απειλή της ακτινοβολίας στην Κεντρική Ασία από τις εξορρυκτικές αυτές δραστηριότητες. Αγαπητέ κύριε Κούκαν, αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής Εξωτερικών, κύριε Νταν Πρέντα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημειώνουμε ότι το ζήτημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης ε, των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις κύριες προτεραιότητές μας. Αναμένουμε λοιπόν την στήριξη των ε, Ευρωβουλευτών και την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την αναλυτική παρουσίασή σας, στην οποία αναφερθήκατε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την χώρα σας και τις ε, σχέσεις της ε, και την επιτυχή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον ε, μόνιμο εισηγητή για την Κυργυζία, τον κύριο Κρίστιαν Νταν Πρέντα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ότι κύριε Υπουργέ. Ε, ακούτε, εντάξει, ακούτε την διερμηνία. Μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία που αναλάβετε να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι μια σημαντική ε, ανταλλαγή απόψεων και επικαιρή γιατί αμέσως μετά θα συζητήσουμε για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι η σύστασή του προς το Συμβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, της ε, Δημοκρατίας της τη αυτής της ε, συνολικής ε, ε, συμφωνίας για την οποία είμαι εισηγητής. Η Κυργιζία ως χώρα της Κεντρικής Ασίας είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που ξεκινάει να παίρνει να, ένα διαφορετικό δρόμο και ήδη από το 2015 είχαμε τα πρώτα ε, σήματα με την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καζακστάν. Ε, έπειτα υπήρξε η εντολή διαπραγμάτευσης προς την ύπατη εκπρόσωπο κ. Μογκερίνη έτσι ώστε να διαπραγματευτεί με ε, μια συμφωνία ενισχυμένη συνεργασίας με το Ουσβεκιστάν και έχουμε ξεκινήσει και διαπραγματεύσεις για μια εταιρική σχέση με το Τουρκμενιστάν. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να ε, ενισχύσει ε, και να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με τις χώρες αυτής της περιοχής επί τη βάση των αναγκών τους από το 2019, όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε μια νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία. Επομένως, είναι προφανές ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μεγάλη πολιτική βούληση έτσι ώστε να ενισχυθεί και να εμβανθυνθεί η συνεργασία με τις χώρες της περιοχής. Θα ήθελα να τονίσω ότι η δημοκρατία της Κυργιζίας είναι χώρα προτεραιότητας για τις σχέσεις μας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Και θα έρθω τώρα και θα μιλήσω πιο λεπτομεριακά για την ε, συμφωνία ε, επί της οποίας έγινε ε, η διαπραγμάτευση και ήδη από την αρχή ως εισηγητής είχα επιμείνει ότι αυτή η συμφωνία θα έπρεπε να ήταν φιλόδοξη. Δηλαδή, μια συμφωνία η οποία θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας, της αγοράς, με τρόπο ο οποίος θα συνεισφέρει στους πολίτες και των δύο μερών και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης η συμφωνία αυτή να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, τους κανόνες του ανταγωνισμού και να ενισχύσει ιδιαίτερα τη διαφάνεια στους ε, θεσμούς. Μια συμφωνία στην οποία θα αναφέρονται και μεγάλα διεθνή προβλήματα όπως το οργανωμένο έγκλημα, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και θα προτείνεται η αντιμετώπιση του στο πλαίσιο της πολυμερούς προσέγγισης. Και θα ήθελα επίσης μια συμφωνία η οποία να ε, προωθεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι η δημοκρατία τη Κυργυζία χώρε η οποία είναι, η οποία είναι μια αναδυόμενη δημοκρατία στην περιοχή. Βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι όλα τέλεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη χώρα σα στο πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Και για να συνεχιστεί αυτό, για να γίνει περισσότερο έντονο αυτό, θέλουμε να υπάρχει και μία δέσμευση από την δική σας την πλευρά σε όλους τους τομεί συμπεριλαμβανομένης και, της, συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με χαροποιεί το γεγονός ότι το άκουσα στην ε, ομιλία σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα επιμείνει στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, στη σημασία που έχει να συζητήσουμε και θέματα σε σχέση με, το δικαστικό σύστημα και την ανεξαρτησία του. Μια έλλειψη ε, διαφάνειας στις δικαστικές διαδικασίες και το σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης. Είναι θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά. Ε, και πριν κλείσω θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία που έχει η ε, εμπάθυνση και η ένταση της περιφερειακής συνεργασίας. Το αναφέρω και στην εκθεσή μου ότι χρειάζεται να λάβουμε όλα τα μέτρα τα απαραίτητα έτσι ώστε να υπάρξει απάλληψη των εντάσεων και των συγκρούσεων που πιθανώ υπάρχουν μεταξύ του Κυριαστάν και των γειτονικών κρατών, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών τη περιοχή για κοινά προβλήματα, όπω για παράδειγμα η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η διαχείριση των υδάτων, η συνεργασία σε αυτούς τους τομείς πιστεύω ότι θα φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ και θα ήθελα να μας ενημερώσετε περισσότερο ε, για αυτό το ζήτημα το τελευταίο ιδιαίτερα, για την περιφερειακή συνεργασία, Ποιε είναι οι εξελίξεις, πώς βλέπετε τη, τη, τις προβλέψεις για το, για το άμεσο μέλλον. ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στη δημοκρατία του Ουσμπεκιστάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων, Άλντε, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας για αυτήν την ε, συμφωνία, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία. γενικώ μιλώντα, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσει την παρουσία τη στην περιοχή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, αυτή η συμφωνία ε, που είναι πολύ θετική, είναι, είναι πολύ θετική και αντίστοιχε συμφωνίε θα πρέπει να γίνουν και με άλλε χώρε τη Κεντρική Ασία. Πιστεύω πως με αυτή τη συμφωνία θα έχουμε μια αποτελεσματικότερη και καλύτερη ακόμα αξιοποίηση αυτών που έχουμε πετύχει στο πλαίσιο της ε, υφιστάμενης ε, ε, συμφωνίας και επίσης θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ στη σημασία που έχει η περιφερειακή συνεργασία, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές στο Ουσμπεκιστάν. Το ανέφερε ήδη και ο συνάδελφος Πρέντα. Πιστεύω ότι ίσως έχουν βελτιωθεί οι πιθανότητες για μια αποτελεσματική συνεργασία. Επίσης, είναι σημαντική η προστασία των μειονοτήτων στο Κυριγιστάν. Γνωρίζετε ότι σε όλες αυτές τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, σε κάθε μια από τις χώρες υπάρχει μια σημαντική μειονότητα από άλλες γειτονικέ χώρες. Ε, ακόμα ένας λόγος για τον οποίο χρειάζεται πιο ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία. Η περιοχή αυτή του κόσμου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, σημαντική από γεωστρατηγική απόψεω. Έχει ε, ε, προσελκύει το ενδιαφέρον τη Ρωσία, τη ε, Κίνα και βλέπουμε εξελίξει. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα πρέπει να βασίζεται στις οικουμενικές αξίες επί των οποίων βασίζεται και η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε εσείς να εκφράζετε αυτές τις αξίες σε αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιο άλλο τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να σχολιάσετε για το ερώτημα το οποίο ετέθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Για το ότι ακριβώς αποδίδεται μεγάλη σημασία στις σχέσεις ε, με την χώρα μου και ακριβώς θέλουμε αμοιβαία υποφελή σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την ε, συμφωνία αυτή που έχουμε συνάψει και θέλουμε και οι δύο πλευρές ε, να ενισχύσουν ε, τους κοινούς δεσμούς μας. Είναι κάτι επί του οποίου εργαζόμαστε Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Ακριβώ προσπαθούμε να συζητήσουμε επικοδομητικά αυτά τα ζητήματα. και να εργαστούμε με τρόπο συντονισμένο, επικοδομητικό για να βρούμε λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. θα ήθελα ακριβώς ε, να ευχαριστήσω και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικοδομητική τους προσέγγιση. Όσον αφορά το σχόλιο, το οποίο έκανε ε, Κροάτης ε, συνάδελφος, θα ήθελα να πω ότι η χώρα μας είναι υπερήφανη για το ότι είναι μια πολυεθνική χώρα, πολυπολιτισμική και με πολλές θρησκείες το ενδιαφέρον βεβαίω ε, και τα συμφέροντα του κάθε πολίτη μας ε, προστατεύονται. Έχουμε πάνω από 80 εθνικότητες ε, στην χώρα μας και κάθε μία από αυτές έχει τα δικαιώματα της τα οποία εγγυάται το Σύνταγμα της χώρας. Όσον αφορά το, στις γλώσσες, έχουν ε, σχολεία στις γλώσσες τους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσει των ε, τοπικών ε, κοινοτήτων και σύμφωνα με το Σύνταγμα έχουμε δύο επίσημες γλώσσες. Η κυργιζική είναι η γλώσσα του κράτους και η γλώσσα επικοινωνίας των διαφόρων εθνοτήτων είναι η ρωσική. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να συναντηθούμε μαζί σας και να ακούσουμε τις ε, απόψεις σας για τις μελλοντικέ ε, σχέσεις ε, μας και ελπίζω να είναι αμοιβαία επωφελής και να ωφελήσουν και την δική σας χώρα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια του μάλλον. Ladies and gentlemen, as you have... Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως θα έχετε διαπιστώσει, τα επόμενα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι ακριβώς θέματα τα οποία αγγίξαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προηγούμενου σημείου. Το μόνο λοιπόν που θα σας πω είναι ότι στις 6 Δεκεμβρίου θα τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά, όπου θα γίνει η ψηφοφορία επί της έκθεσης α, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία η τελική. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Πρόκειται για δημόσια ακρόαση για τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη σχέση μας με τη Ρωσία, πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουμε την σημασία που έχει να συνεχίσετε ανοιχτός ο διάλογος με τη Ρωσία, ενώ βέβαια παραμένουμε πιστοί και στις αξίες μας. Αυτός ο διάλογος ε, έχει εξεταστεί από το, την κυρία Κανιέτε στη έκθεσή της για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, την οποία θα συζητήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω δύο ε, ειδικού στα θέματα της Ρωσίας και των ε, σχέσεων μετά την Σοβιετική Ένωση, των πολιτικών σχέσεων, την κυρία Μεντράς από το, την Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι και θα συζητήσουμε για το μέλλον αυτών των σχέσεων ε, με την κυρία Μετράς και τον κύριο Σφέστσικ ε, για τις σχέσεις μας λοιπόν και το μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. θα ακούσουμε διαδοχικά τις ε, δύο ειδικού τις δύο εμπειρογνώμονες. Έχετε το λόγο κύριε Μετράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερο ευτυχή που επιστρέφω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι το, εκείνο το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει αποδείξει ότι συστηματικά και συνεκτικά αντιλαμβάνεται τη σημασία της Ρωσίας και τη σημασία της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτούς τους κοινούς μας γείτονες της, τη, τη Ρωσία και με την ίδια τη Ρωσία αλλά και με τις χώρες που βρίσκονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία γεωγραφικά εννοώ. Και μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία από το 2014 είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί κανείς να συζητά τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνει συστάσεις προς την Ουκρανία χωρίς να λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα και την σχέση της Ρωσίας με την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Μου ζητήθηκε να ξεκινήσω την παρουσίασή μου από τις πέντε αρχές του 2016 που περιγράφονται στα συμπεράσματα των 28 Υπουργών Εξωτερικών και τις οποίες έχει ενστερνιστεί και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το ερώτημα βέβαια είναι τι πρέπει να γίνει στο μέλλον από το 2019-2021. Θα προσπαθήσω να το πράξω αυτό όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Και είμαι σίγουρη ότι τα ζητήματα αυτά θα τα συζητήσουμε και ευρύτερα. Το βασικό επιχείρημα που θέλω να σας παρουσιάσω είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς μεγάλες προκλήσεις, αλλά η Ρωσία και η ρωσική κοινωνία και η ουκρανική κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Το συμπέρασμα αυτής της διαπίστωσης είναι ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε στη διάθεσή μας πολύ περισσότερα εργαλεία για να βρούμε λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις από ό,τι οι αρχές της Ρωσίας. Και αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε, να εξηγήσουμε, να δημοσιοποιήσουμε στην, στους πολίτες μας και στις κυβερνήσεις μας. Ότι έχουμε στα χέρια μας δηλαδή πολύ καλύτερα εργαλεία. Ξεκινώ λοιπόν από αυτές τις πέντε αρχές του 2016. Οι πρώτες τρεις έχουν ουσιαστικά σχέση με τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Δηλαδή, ζητήθηκε να γίνει πλήρης εφαρμογή τη συμφωνία του Μίνσκ και ότι θα διατηρηθούν οι κυρώσει μέχρι να συμβεί αυτό. Δεύτερον, ζητήθηκε να υπάρξουν ε, στενότερε σχέσει με τι πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίες και τρίτον, να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε πιθανέ απειλέ από τη Ρουσία όσον αφορά την ενέργεια, το ίντερνετ, ε, την παραπληροφόρηση κτλ. Θα έλεγα ότι η εφαρμογή αυτών των τριών αρχών έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και στα 28 κράτη-μέλη, ακόμα και σε εκείνες τις λεγόμενες ανελεύθερες, αν θέλετε, κυβερνήσεις, ορισμένες κυβερνήσεις οι οποίες έχουν δείξει τέτοιες τάσεις εντός της Ένωσης. Θα έλεγα ότι ακολουθούμε αυτές τις τρεις αρχές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτές οι τρεις αρχές δεν συνιστούν πολιτική. Δεν αρκούν για να έχει κανείς πολιτική και αυτό είναι το πρόβλημά μας, γιατί αν δούμε τις επόμενες δύο, θα γελάσετε. Λένε οι επόμενε δύο. Παρά τι εντάσει να εμπλακούμε και να συνεργαστούμε με τη Ρωσία για την Μέση Ανατολή, τον, την τρομοκρατία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και η πέμπτη αρχή είναι να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς τον κοινωνία των πολιτών, δηλαδή αυτό που υποτίθεται ότι κάνουμε εδώ και δεκαετίε από το 1990 και μετά. Οι αρχέ ε, θεωρητικά είναι σωστές, Υπάρχει η πολιτική βούληση και υπάρχει η οικονομική βούληση σε ένα βαθμό, υποστηρίζουμε την Ουκρανία για παράδειγμα, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τη και την αντιμετώπιση των επίγουσων καταστάσεων και των βραχυπρόθεσμων και μέσοπρόθεσμων δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει. Και ελπίζω να καταφέρουμε να συνεργαστούμε ε, και να καταλήξουμε σε ε, μια έκθεση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας η οποία να περιέχει πολύ περισσότερες προτάσεις από ότι άσκηση κριτικής. Πρέπει να ανανεώσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξετάσουμε σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία τρία χρόνια στο πολιτικό πλαίσιο. Από τότε δηλαδή που υιοθετήθηκαν αυτές οι πέντε αρχές και αντιστοίχως να προσαρμοστούμε. Αλλαγές από το 2016. Η κατάσταση στην Κρυμαία έχει επιδεινωθεί. Στον Τον και ε, είναι, είναι, ήταν λογικό, δεν θα μπορούσε παρά να πάει προς το χειρότερο. Ε, είναι μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει σεβασμός του νόμου, υπάρχουν δολοφονίες, υπάρχουν παράνομες εκλογές, υπάρχουν παράνομοι κυβερνήτες. Και με λύπη μου διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα και βουλευτές ή πρώην βουλευτές από τις χώρες μας, οι, οποίοι επισκέφτηκαν τον Τόνιενσκ για να λειτουργήσουν ω παρατηρητές αυτών των παράνομων εκλογών. Κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να το είχαμε καταγγείλει. Το Κίεβο ε, έχει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για να καταρτήσει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του στο, στο Ντόνενσκ και αλλού. Επομένως, η συμφωνία του Μίνσκ καταραίει. Είναι εύκολο αν κάποιο θέλει να ασκήσει κριτική στη συμφωνία του Μίνσκ να, Μίνσκ, να πει δεν λειτουργεί. Ε, Βεβαίω εφαρμόζουμε τι κυρώσει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχω επισκεφτεί την Ουκρανία και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η κυρία Χάρμς, την έχουν επισκεφτεί την Ουκρανία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προτείνουμε νέες πολιτικές έτσι ώστε να βοηθήσουμε το Κίεβο να παραμείνει σε επαφή με τους πολίτες τους Ουκρανούς που παραμένουν στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη. Δεύτερη αλλαγή. Ο πόλεμος στη Συρία. Το 2016 υπήρχαν ακόμα ορισμένοι ειδικοί, ορισμένες κυβερνήσεις οι οποίοι πίστευαν ότι θα μπορούσε θεωρητικά κάποια στιγμή να παίξει ένα θετικό ρόλο η Ρωσία. Αν όχι να αναλάβει μια ε, συμμετοχή στη στρατιωτική σύγκρουση, δεν ήταν αυτό ο στόχος, αλλά τουλάχιστον να βοηθήσει στην έξοδο από τη σύγκρουση. Καταρχήν, ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονό ότι στην αρχή η Ρωσία υποστήριξε το καστός του Αλάσαντ ε, και τώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη και βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Βασιστήκαμε σε μία παγκόσμια δύναμη όπως η Ρωσία, δεν λειτουργήσε αυτή η ε, αναμονή και το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εμπλακεί, θα προσπαθήσει να ανεκοδομήσει τη Συρία χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα για το ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας και τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Τρίτο θέμα. Μετανάστευση σε σχέση πάλι με το προσφυγικό. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Έχει εξελιχθεί από το 2016, επιδεινώθηκε το 2017 και συνεχίζει. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν βοηθά σε αυτό το τομέα γιατί η Ρωσία συνεχίζει να υποστηρίζει παραπληροφόρηση και τέτοιες εκστρατείες. Και οπωσδήποτε έχει έναν ρόλο στην επιδείνωση αυτού του οποίου λέμε λαϊκισμός, ε, ξενοφοβία Τέσσερις ε, μεγάλες αλλαγές. Η ρωσική ηγεσία και η ελίτ ε, που κυβερνά συμπεριφέρονται πλέον σαν να βρίσκονται υπό πολυερκία. Δεν ακούνε το λαό τους, δεν ακούν τις διαμαρτυρίες, η οικονομία ε, εξακολουθεί να επιβραδύνεται και η καταστολή αυξάνεται. Αλλά αυξάνονται και οι διαμαρτυρίες. το οποίο σημαίνει ότι στην παραδοσιακή πολιτική που έχουμε τη στήριξη κοινωνία των πολιτών πρέπει να ξαναδούμε τις μεθόδους μας. Πρέπει να σκεφτούμε την Ρωσία ως μια χώρα με κοινωνία, όχι μόνο κοινωνία των πολιτών, ακτιβιστές ε, στις μεγάλες πόλεις ε, που μιλάνε αγγλικά και έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Ας σκεφτούμε τη Ρωσία ως μια φυσιολογική κοινωνία, όπως ε, εμείς. Γιατί και η Ουκρανία ε, σημειώνει πρόοδο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα όταν μιλάμε για δημοκρατία και κράτος δικαίου, λογοδοσία και εναλλαγή. Δηλαδή αυτοί που έχουν την εξουσία είναι προσωρινοί, δεν είναι ιδιοκτήτε, Οπότε ας παρακολουθήσουμε στενά το τι συμβαίνει προσεκτικά στη Ρωσία, όχι μόνο στη Ρωσία, στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη έχουμε πολλούς ειδικού ε, Ρώσους, Ευρωπαίους, Ουκρανούς. Ε. ε, ας τους ακούσουμε λοιπόν ε, και θα μας πούν πολλά. Μια με άλλη μεγάλη αλλαγή Ε, και βέβαια ε, αλλάζουν οι γειτονιέ. Ε, η Αρμενία, η Ουκρανία, υπάρχει μια ακτίδα ελπίδας στην Γεωργία. Όλες αυτές οι τάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας δείχνουν μια αργή εξαφάνιση της σφαίρας επιρροής της Μόσχας. Γιατί η Μόσχα πλέον δεν είναι ελκυστική για τις νέες κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Υπάρχει επίσης σε αυτήν την φάση κάτι το οποίο ακούω ήδη ε, τους επιφυλακτικούς να λένε «Α, ναι, αλλά να ακούσουμε εσάς ε, και κάνουμε κάτι όπως αυτό που λέτε θα έρθουμε σε σύγκρουση με τη Μόσχα». και η Μόσχα είναι σημαντικός τα λοιπά. Το παίρνω στο σοβαρά. Εγώ θα πάω στη Μόσχα τη Δευτέρα και θα μιλήσω σε όσους θέλουν να μου μιλήσουν. Και θα απαντούσα ως εξής. Ε, από το 2014 η ηγεσία του Πούτιν μας είχε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν ήθελε να συζητήσει μαζί μα τα ζητήματα της ασφάλειας. Και όχι μόνο τη στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και την ε, ανθρώπινη ασφάλεια του λαού. Η δεύτερη μου απάντηση είναι δυστυχώς ότι έχω παρατηρήσει το καθεστώς στη Μόσχα να μου λέει ότι ό,τι κάνουμε αν ε, το γλυκάνουμε λίγο το χάπι θα τους ανταγωνιστούμε γιατί το πρόβλημα δεν είναι δικό μας είναι δικό τους εσωτερικό των ρωσικών ελίτ που ανησυχούν όλο και περισσότερο και αισθάνονται υπό πολιορκία και καταλήγοντας ε, θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική για το τι είχαμε κάνει στο παρελθόν. Ε, και, αλλά πρέπει να συγχαρούμε και αυτούς, ε, καλό είναι αυτό, έτσι, ψυχοφελές. Και να κάνουμε κάποιες ομάδες συνομιλιών, όπως κάνουμε εδώ πέρα, στο εκτελεστικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά είμαι σίγουρη ότι νέες ιδέες ε, και νέες μορφές ε, επαφών ε, λειτουργούν. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ένα θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι τόσο μεγάλο σημείο αναφορά στη Ρωσία για όλους. Όλοι γνωρίζουν την απόφαση για τον Αλεξέη Ναβάλνη. Δηλαδή μόνο το ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητο δικαστήριο που δεν είναι εθνικό αλλά συλλογικό είναι ένα σημείο αναφοράς ε, για αυτούς ε, στην Ρωσία που θέλουν να παραμείνουν εκεί, να δουλέψουν για τη χώρα τους ε, και να τα πάνε καλύτερα. Χωρίς να πάνε στην φυλακή. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε και περισσότερες συζητήσεις και προτάσεις ε, ε, και λυπούμε όμως γιατί μετά θα πρέπει να φύγω να πάω στο Μιντι γιατί έχω μάθημα να κάνω στο Παρίσι στις 2.30 ε, ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι δημόσια διοίκηση και ο συνάδελφος Στρεβίσιους έχει ζητήσει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το προνόμιο να μιλήσω πρώτος. Μπορώ να συμφωνήσω ότι οι αρχές που επεξεργαστήκαμε μετά από τον Ρωσικό πόλεμο στην ε, ε, Ουκρανία είναι ε, κατά κάποιο τρόπο εμβολιασμό της δύση κατά του αντικτύπου και της επιρροής της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουμε προσκολλημένοι στις αρχές αυτές. Αλλά δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κάποιος ε, ε, που να αμφισβητεί αυτές τις αρχές από τη δυτική πλευρά. Ο κύριος Σαλβίνη το κάνει πάρα πολύ καλά και είναι μάλιστα, έχει την εξουσία ε, και εκπροσωπεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα ας μην είμαστε και τόσο αισιόδοξοι γίνονται προσπάθειες αμφισβήτησης και ενδεχομένως αναθεώρησης ε, αυτής της πορείας. Η θέση σας ότι η επιρροή της Ρωσίας ε, στην ε, γειτονιά της μειώνεται. Ναι, ίσως στους πολύ κοντινούς γείτονες, γιατί δεν υπάρχει θετικός αντίκτυπος. Λίγα μπορούν να πουλήσουν οι Ρώσοι στους γειτόνους τους. Άρα άμεση πίεση ε, ή παρεμβατικά μέτρα, ας πούμε. Ναι, αλλά και πάλι ας μην κλείνουμε τα μάτια μας όσον αφορά αυτό το outreach, αυτή την προσπάθεια προσέγγισης. Μεγαλύτερη προσπάθεια προσέγγισης βέβαια γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, πέρα από τους κοντινούς γείτονες. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά να ασκούν την αρχή «Διέρη και Βασίλευε». Η, Ευρω... η Ρωσία δεν θέλει ευρωμένη Ευρώπη. Δεν μιλάει για το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα project, ένα σχέδιο ειρήνης, ανάπτυξης κλπ. Απλώς προσπαθούν να μας διαιρέσουν και θέλουν να ε, ε, μας κατεβάσουν στο επίπεδο κρατών εθνών. Εδώ πρόκειται για πραγματική ε, παράβαση της αρχής της ΕΕ και μπορεί να λειτουργήσει ε, η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχει άμεση αντιστοίχηση ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την θέση του προπολογισμού αυτών των δύο στοιχείων. Ε, εμείς διαρκώς λέμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω της κλιματικής αλλαγής για να μειώσουμε την επιρροή της Ρωσίας. 14, ε, στην περίοδο 14-18 αυτό που ανέπτυξε η Ρωσία είναι τα fake news και η παραπληροφόρηση και η επιρροή που μπορεί να έχουν αυτά σε μας. Μήπως θα μπορούσατε να εξειδικεύσετε λίγο σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για αυτή την κατάσταση. Όταν ε, θα πάτε στη Μόσχα, αν ρωτήσετε ε, ε, είναι η Ρωσία πίσω από αυτά, ε, ή αν ρωτήσετε ας πούμε κάποιον υπεύθυνο υπάρχει κάποιος αξιωματούχος Ρώσος πίσω από τα fake news που έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, οπωσδήποτε θα πέσετε πάνω σε ένα τείχο άρνησης και ο κ. Σουκόφ ε, και οι υπόλοιποι οπωσδήποτε θα ξεγλιστρήσουν από τον διάλογο αυτό. Και τελικά εμείς οι ίδιοι κάνουμε το διάλογο μεταξύ μας. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ποια είναι η άποψή σα, λοιπόν όσον αφορά τα fake news, ψευδεί ειδήσει και παραπληροφόρηση. Ποια είναι η εκτίμησή σα πώς αξιολογείτε τη θέση και ποια θα πρέπει κατά την άποψή σας να είναι η θέση της Ευρώπης. Τι μπορεί να δώσει αποτελέσματα και τι όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι τώρα προς την Σάντρα Καλνιέτε, την εισηγήτρια παρακαλώ. Δεν ζήτησε το λόγο, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να μιλήσεις. Εγώ θα κάνω και τις ε, τελικές παρατηρήσεις στο τέλος, συμπερασματικέ. αλλά, αλλά πραγματικά ε, θα αφήσω το λόγο στους συναδέλφους που ξέρουν καλά το θέμα και είναι εμπειρογνώμονες. Βεβαίω ξέρω ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι που είναι persona non grata στη Ρωσία. Θα ακούσω λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικά. Σε άκουσα κυρία Μεντρέσε, σας άκουσα πολύ προσεκτικά Μαρή Μεντρέσε. Θα ακούσω και προσεκτικά όλους όσους, ε, όσοι μιλήσουν και εσάς ε, και μετά ε, θα, θα κάνω εγώ τα συμπερασματικά σχόλια. Ο κύριος Γιούρεκ, θα μιλήσω στα πολωνικά εγώ. Αν θέλετε λοιπόν βάλτε τα ακουστικά σας για να καταλάβετε τι σας λέω. E, e, Ευχαριστώ. Η Ρωσία απειλεί πρώτα απ' όλα τους γειτονές της ε, και ε, είναι μια περιφερειακή απειλή. Απειλεί τους γείτονές της ε, και όλοι γνωρίζουμε το δόγμα του ρωσικού κράτους ε, που θεωρεί το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης ως μια μεγάλη καταστροφή και θέλει να δημιουργήσει μια ρωσική σφαίρα επιρροής. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και συχνά το βλέπουμε επιφανειακά μόνο χάρη. Όταν έχουμε Γεωργιανούς εδώ, μιλάμε για τα κατεχόμενα της Γεωργίας, όταν δεν είναι εδώ δεν μιλάμε κανείς. Διαμαρτυρόμαστε για την Κρυμαία, αλλά το πιο αποτελεσματικό θα ήταν να αποκαταστήσουμε την στρατηγική ισορροπία. Όποτε χειροτερεύει η κατάσταση στην Ρωσία θα έπρεπε να μειώνει την ασφάλεια της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα τέτοιο. Η Γεωργία και η Ουκρανία δεν ε, μας απασχολούν τόσο όσο πριν από λίγα χρόνια και όπως είπε η καθηγήτρια, παρά τις ε, συμφωνίες, η κατάσταση στην Κρυμαία επιδεινώνεται. Αντί να εμπλεκόμαστε, να ζητούμε κάποιες ε, προκλήσεις ε, περιτές ε, και λέμε εντάξει η Ρωσία πολεμάει στο πλευρό του Άσαντ. Η άλλη πλευρά ποια είναι όμως η Ρεία, η και οι φονταμενταλιστές που συνδέονται με το ISIS. Είναι μια τεράστια τραγωδία και δεν θα υπήρχε εμπλοκή της Ρωσίας εάν ε, δεν είχε παραταθεί αχρίαστα αυτός ο πόλεμος τόσα χρόνια. Το χειρότερο δε είναι τα ρωσικά επιχειρήματα για τις εσωτερικές ε, πολιτικές συγκρούσεις όταν μιλάμε για ενίσχυση εθνικιστικών λαϊκιστικών ε, ρευμάτων. Έχω μία πάρα πολύ απλή πρόταση. Αν σταματήσουμε να αποκλείουμε πολιτικά εκατομμύρια Ευρωπαίους, ε, τότε θα σταματήσει και η ρωσική επιρροή στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματική ασφάλεια. Και βεβαίως ε, συχνά μιλάμε για αυτό το τρομερό αυταρχικό καθεστώς ε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, είναι ένα σημαντικός εταίρος και το Μεκεβέλη και τα λοιπά. Τόσα λέει δηλαδή. Οπότε ας εστιάσουμε στην ασφαλειά μας, στο να υπερασπίσουμε τις χώρες μας και να μην αναζητούμε εσωτερικούς εχθρούς. Θα απελευθερώσουμε τον κόσμο από την ρωσική προϊόντα όταν αρχίσουμε να σεβόμαστε αλλήλους. Σας ευχαριστώ κύριε Γιούρα. Κάλους δύο μιλητές έχω. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, η κυρία καθηγήτρια έχει να διδάξει το απόγευμα στο Παρίσι, οπότε σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο. Ε, βεβαίως, ε, αφού απαντήσει θα αφήσει εδώ τον κύριο Σεύτσικ, ε, τον οποίον επίσης μπορούμε να ακούσουμε. Κύριος Χατζηγεωργίου. Good Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Μία ερώτηση έχω μόνο, η οποία σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φαίνεται ε, απλή, αλλά είναι σε δεύτερη ανάγνωση βαθιά πολιτική. Ε, ε, διαφορά ανάμεσα στον Πατριάρχη της ε, ε, Ρωσίας και του της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την Αρχιεπισκοπή της Ουκρανίας. Εκεί αφορά η ερώτησή μου. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθαρά θρησκευτικό το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να επανασυνδέσει με κάποιες σχέσεις της με την Συρία, την Αντιοχία κλπ. Κάποιες άλλες δηλαδή εκκλησίες εις την Ανατολή. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δυο πάνω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το 2016 είχαμε ένα ψήφισμα σχετικά με την στρατηγική επικοινωνιακή ατζέντα της Ένωσης για τη Ρωσία. Χθες εδώ στην Επιτροπή μας, δύο χρόνια μετά, συζητήσαμε την εξέλιξη της κατάστασης και τι μπορούμε να κάνουμε και χαίρομαι γιατί ε, είναι περισσότερες οι πολιτικές ομάδες οι οποίες υποστηρίζουν αυτό το θέμα που αποτελεί απειλή και για μας, για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και αυτό που είπε ο Πίτερ Αστροβίσιος, ε, συμφωνώ μαζί του, δηλαδή ερώτηση πώς μπορεί κατά την άποψή σας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την προπαγάνδα. Δεύτερο ερώτημα, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πολλοί μεταξύ ημών ε, ε, παρουσιαζόμαστε ως ρωσόφοβοι. Ε, είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει ρωσοφοβία και δεν είναι ο κόσμος ρωσοφοβικός. Ε, ε, ε, ξέρουμε, αγαπάμε τη Ρωσία, την πατρίδα του Τσαϊκόφσκι, του Ροστροπόφ. δεν έχει καμία σχέση αυτό με το τι συμβαίνει στη χώρα και το τι κάνει η πολιτική ελίτ η οποία ε, ζει κατά τον δυτικό τρόπο ζωής, ε, ε, στέλνει τις οικογένειές τους να ζήσουν στην Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν με λαϊκίστικο τρόπο την πολιτική και τη ζωή στην Ευρώπη. Την Ρωσία την αγαπάμε, το λέω και το υπογραμμίζω, καμία σχέση δεν έχουν αυτά. Τελευταία, τελευταία η ομιλήτρια, η κυρία Γιάκονσάρη. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι πολύ σύντομη. Κυρία Μεντράς, είπατε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ίσως ε, θα πρέπει να ασκήσουμε αυτοκριτική. Ποιο είναι το λάθος που κάναμε στις σχέσεις μας με την ε, Ρωσία και ποια είναι τα λάθη τα οποία ε, εξακολουθούμε ενδεχομένως να κάνουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι κακή για όλους, lose-lose situation. Ποιοι ε, ε, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο αυτής της αυτοκριτικής. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μανδράς, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη, γιατί μην λησμονούμε ότι έχουμε άλλον έναν ε, ομιλητή προβλέψει και ελπίζω, αγαπητέ συνάδελφοι, ότι θα με βοηθήσεις λίγο στην απάντηση που θα πρέπει να, ή στις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσω σχετικά με το ερώτημα του πρώτου ομιλητή. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί αυτό αφορά το δεύτερο τμήμα της ε, παρέμβασής μου και δεν, το, δεν κατάφερα να το αναπτύξω γιατί έπρεπε να είμαι σύντομη. Όλα αυτά που λέτε ισχύουν, είναι σωστά αλλά ίσως να διαφωνήσουμε ελαφρά σε ένα σημείο, σχετικά δηλαδή με, την, με τις διασυνδέσεις, ε, τις correlations. Όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία αναφέρατε ισχύουν, είναι αληθή. Το πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο τα αναλύομαι και τα ερμηνεύομαι. Πώς αναλύομαι και ερμηνεύομαι την, το συσχετισμό ανάμεσα, ας πούμε, στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και τη θέση του κυρίου Σαλβίνη στην Ιταλία ή πώς διασυνδέουμε την μετανάστευση και την πληροφόρηση για τις ε, μεταναστευτικές ροές και την νίκη ε, της, του συνασπισμού Σαλβίνη πέντε αστέρες στην Ιταλία. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και στην Ισπανία. Πιστεύω ότι αυτά είναι κεντρικά στοιχεία για σας ως ευρωβουλευτές. Δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούμε να διασυνδέσουμε, να συσχετίσουμε φιλόδοξες ευρωπαϊκές πολιτικές με λογικές, συνεκτικές και υποστηρικτικές πολιτικές ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί οι κύριες εκλογές θα πρέπει να ε, να ε, κερδιθούν από πλειοψηφία φιλοευρωπαϊκών κομμάτων. Αυτό έχουμε κατά νου όλοι. Άρα πρέπει ε, οι δημόσιες σχέσεις μας, τα PR, να βελτιωθούν και η επικοινωνία και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι όχι. Ο κόσμος δεν ασθενεί βαρέως λόγω μιας ε, νέας ε, λιμόδους ε, νόσου που περιδιαβαίνει την Ευρώπη από την Πολωνία στην Ιταλία και Τούμπαλιν ε, και ζητώ συγγνώμη τους Πολωνούς φίλους, αλλά ε, που αναφέρομαι στην, ε, στις κυβερνήσεις Πολωνίας ή της Ουγγαρίας. Όχι, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Υπάρχουν παρόμοια συμπτώματα σε πολλές χώρες, συχνότερα από παλιότερα ίσως. Αλλά ε, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε για την Πολωνία, είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα εντός τους. Russia... Ε, εγώ διαβάζω λίγο τον υποτιτλισμό αυτών που είπατε. Ε, είναι ισχυρή η Ρωσία, είναι ισχυρός ο στρατός της και θέλουν ε, να προελάβουν. Όχι, όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν μια τέτοια άποψη. Δεν, ε, στο Νταμπάς δεν πήγαν ως ε, ε, κατακτητές, στην Συρία δεν πήγαν ως κατακτητές. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό. και βεβαίως στην ε, Ρωσία δεν πηγαίνω για να ε, ε, βρω πραγματικά περιστατικά, αλλά για να μου μεταλαμπαδεύσουν τη σοφία τους οι φίλοι και οι γνώστες που ζουν εκεί. Γιατί αυτοί μου λένε ότι και εμείς οι διανοητές που, και οι διανοούμενοι μάλλον που ακούμε και αγγλικά μέσα ενημέρωσης ή μάλλον μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά, δεν επηρεαζόμαστε ε, ε, από αυτά που λένε τα δικά μας ρώσικα μέσα, αλλά αυτά που λένε τα δικά σας ε, δυτικά μέσα περί ασθενείας και περί αποδυνάμωσης της Ευρώπης κλπ. Επομένω, επομένως, όσον αφορά την παραπληροφόρηση, όλες οι πλευρές θα πρέπει να καταπολεμήσουν την ε, παραπληροφόρηση και νομίζω ότι από πλευράς τη Ευρωπαϊκής Ένωση όντω το δουλεύουμε πολύ, πρέπει να το δουλέψουμε και περισσότερο και οπωσδήποτε θα πρέπει εμείς να οικοδομήσουμε το δικό μας αφήγημα ή τα δικά μας αφηγήματα και να προωθήσουμε τα καλά νέα, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε πολλά καλά νέα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ε, ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι είναι ευτυχής ο κόσμος που ζει στην Ευρώπη. Το θέμα για την ε, Πολωνία θα το αφήσω στον Μπάρτ. Θα ήθελα μονάχα να υπογραμμίσω ότι ήμουν ιδιαίτερος ευτυχής ε, που μοιράστηκα ε, την χαρά των 100 χρόνων από την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Όπως γνωρίζετε πάντως, όλες οι χώρες οι οποίες ανέκτησαν την κυριαρχία τους στην Ευρώπη 100 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, χτες ή προχτές ή παλιότερα, όλες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η ακαιρεότητα είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να μοιραστούν. Δεν θέλουν να μοιραστούν την κυριαρχία και την... Ε, αυτοί που δεν θέλουν να συμμοιραστούν την κυριαρχία τους ή την άμυνά τους δεν θα έχουν πολύ ε, ε φωτεινό μέλλον και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ε, ασφάλεια. Η πραγματική ασφάλεια, η αληθινή ασφάλεια είναι η ασφάλεια των ατόμων και η ύπαρξη θεσμών που μπορούν να προστατεύσουν τα άτομα αυτά. Η αληθινή ασφάλεια είναι είναι αυτή η ασφάλεια που δίνουν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά για να επιτευχθεί αυτή η ασφάλεια θα πρέπει να νοιαστείτε πρώτα για την ασφάλεια των γειτόνων σας, γιατί τα σύνορα έχουν χάσει την παραδοσιακή δομή των σύνορων. Οι Τινήσοι, οι Ουκρανοί, οι πολίτες της Γεωργίας, ε, κινούνται, μετακινούνται. Δεν υπάρχει η έννοια της ασφάλειας η οποία θα περιορίζεται από την ε, συσταλτική έννοια της ασφάλειας εντός των συνόρων μιας χώρας. Η πραγματική ασφάλεια λοιπόν ε, πρέπει να είναι πλέον μια ευρία αντίληψη και οπωσδήποτε μια πιο περίπλοκη αντίληψη της ασφάλειας. ίσως ε, και την τελική ερώτηση, δηλαδή σχετικά με το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, θα το επαναλάβω. Δεν είναι μιλάμε για στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά στήριξη των δημοκρατικών θεσμών, των δημοκρατικών οργανισμών, την, ε, ε, την πολιτική, την χάραξη στρατηγικής κλπ. Πολλοί τρόποι μπορούν να μας Μέσω πολλών ε, τρόπων ε, μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και ε, ευελπιστώ ότι μπορώ να σας βοηθήσω κυρία Βουλευτά για να, στην έκθεσή σας. Κοιτάξτε, εδώ και 40 χρόνια πηγαίνω στη χώρα αυτή και αυτό βεβαίως γίνεται γιατί την αγαπώ πολύ. Αλλά φυσικά οι ελίτ που βρίσκονται στο τιμόνι της χώρας με αφήνουν λίγο με περίπλοκα συναισθήματα. Όσον αφορά το τελευταίο ε, σχόλιο για μια κατάσταση ε, κακή για όλους, lose-lose situation, εγώ δεν το βλέπω έτσι, καθόλου μάλιστα. το 2014 η αλληλεγγύη που δείξαμε και η ισχυρή ε, απόφαση ναι όντως εξέπληξε λίγο την Ρωσία. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι αφήσαμε ποτέ την κατάσταση να φτάσει σε μια lose-lose situation. Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου, δεν ακούνε οι Δεν ε, συμμερίζομαι την άποψή σας, αλλά νομίζω ότι ο Μπάρτ ε, είναι καλύτερα να απαντήσει και να προσπαθήσει να σας πείσει. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ που με ακούσατε. Madam Professor, thank you very much indeed for coming, sharing. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και μοιραστήκατε τις απόψεις σας ε, μαζί μας. Ε, ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Συνεχίζουμε τώρα. Μια που είναι εδώ πέρα ο κύριος Σεύτσικ. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που δεν έχουν καλυφθεί, οπότε έχετε περιθώριο να μιλήσετε, αλλά δεδομένου του χρόνου θα ήθελα να μας πείτε τα βασικά. Και να αφήσουμε και περιθώριο για να κάνουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Ισίτα. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα. Είμαι σύμβουλος ε, στο Think Tank της Κομισιόν, αλλά οι απόψεις που θα εκφράσω είναι προσωπικές. Διδάσκω Βεβαίω, ε, και στο Σιάνσπο, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα εστιαστώ στις μεσοπρόθεσμε ε, προκλήσεις ε, που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για την Ευρώπη και την ευρύτερη φιλελεύθερη τάξη. Πρώτα απ' όλα όμως να θέσουμε τις σχέσεις στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. αυτό το οποίο έχουμε ως γενικότερο υπόδειγμα είναι ο ανταγωνισμός των μεγάλων ε, δυνάμεων και έχει ξανά επανέλθει ο ανταγωνισμός μεταξύ δημοκρατιών και αυταρχικών καθιστώτων μετά από 25 χρόνια συνένεσης. Αν το σκεφτείτε, σχεδόν από το 1989 οι σχέσεις μεταξύ η Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν συνενετικές και είχαν περιγραφεί ως μια κοινωνικοπολιτική σύγκληση και η Ρωσία θεωρούταν ως μια πιθανή υποψήφια χώρα. Βεβαίω υπήρχαν διάφορε συγκρούσει όπω η εισβολή του ΝΑΤΟ στο Κοσφοπέδιο και τη Ρωσία ε, στην Γεωργία, αλλά γενικότερα υπήρχε μια διάθεση συνεργασία και η Ρωσία συνένεσε στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ρωσία μπήκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η G7 έγιναν G8, έγινε δεκτή στον ΠΟΕ, υπήρξε νέα συνθήκη μείωση των στρατηγικών όπλων ε, και συμφώνησε ο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβει τον ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Παρόλε τις ε, διαφωνίες, ε, το 2014 ήταν σαφώς ένα σημείο καμπής αυτό σήμαινε μια σαφή παραβίαση της διεθνούς τάξης και ακολούθησε η παρέμβαση στην Συρία με στρατό και εξοπλισμό του 2015. Και είχαμε ακριβώς ε, την επιδείνωση της διαδικασίας στην χώρα αυτή. Η εκλογική διαδικασία το 16 και το 17 στην Ρωσία επίσης ε, οδήγησε μια κλιμάκωση που δεν είχαμε δει από το τέλος ε, του ψυχρού πολέμου. Μία από τις κύριες προκλήσεις λοιπόν ε, προς την Ευρώπη θα συνεχίσει να προέρχεται από την Ρωσία. Επίσης το ότι χρησιμοποιήθηκαν βιολογικά όπλα στο Ηνωμένο Βασίλειο για δολοφονία ενός κατασκόπου είναι άλλο ένα σημείο κλιμάκωσης. Βεβαίως συχνά ιστορικά λέμε ότι η πρόκληση προέρχεται από τις ανερχόμενες ε, δυνάμεις. Ε, στην περίπτωση της Ρωσίας είναι η στασιμότητα αυτή η οποία δημιουργεί το πρόβλημα ως ε, ένας supernova. Σε γενικές γραμμές η Ρωσία έχει παραμείνει στάσιμη όσον αφορά το υλικό πεδίο τα τελευταία 25 χρόνια. Ο πληθυσμός της έχει μειωθεί και το ΑΕΠ κατά είναι οριακά σήμερα α, μεγαλύτερο σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την οικονομία της. Είναι λοιπόν μάλλον όχι μια μεγάλη δύναμη, αλλά μια περιφερειακή δύναμη. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να φέρεται όσο μεγάλη δύναμη και θεωρείται τέτοια επενδύει στον στρατό τη και οι δαπάνε ε, αυξήθηκαν μεταξύ 2011 και 2016 με 10% ετησίω ε, και ε, είναι γύρω στο 4% του ΑΕΠ, 3% στη ΣΥΠΑ και 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο. Βεβαίως οι δαπάνε αυτέ δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται και θα πρέπει να επανελθεί στον ιστορικό μέσο όρο η Ρωσία. Τώρα, μία από τι βασικέ επιτυχίε ε, τη στρατηγική τη Ένωσης προ την Ρωσία είναι οι κυρώσει. Και εάν δείτε τον αντίκτυπο των κυρώσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κυρώσεις, ε, η ΙΠΑ, Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία έχουν επιβάλει ένα κόστος 1-1,5% ε, του ρωσικού ΑΕΠ ε, πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή από το 2014. Και οι κυρώσεις αυτές φαίνεται ότι πετυχαίνουν να περιορίσουν τις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας. Η οικονομική πίεση στη Ρωσία οδήγησε μείωση του ΑΕΠ το 2015 και 2016 και την ανάγκασε να μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 20% το 2017. Σε αντίση με αυτό, μεταξύ 2000 και 2014 οι στρατιωτικές δαπάνες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, 8% κάθε χρόνο αυξανόταν. Παρά το ότι το Κρεμλίνο δεν έχει αλλάξει την επιθετική του στάση και τον τελικό του στόχο να και δεν έχουμε καταφέρει να αναγκάσουμε το Κρεμλίνο να τερματίσει την ε, σύγκρουση στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η στρατηγική μας για να περισφίξουμε την Ρωσία ως ένας άλλος πίθωνας αποδίδει. Τώρα, ο ρόλος ε, της Ρωσίας συχνά είναι αποσταθεροποιητικός. Στην Ουκρανία προσπάθησε να διασπείρει το χάος ε, και να πνίξει την δημοκρατία με το να αρπάξει δια της βίας την ε, Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία. Τα ρωσικά όνειρα περί Νέας Ρωσίας απειλούσαν να κατακαιρματίσουν περαιτέρω την Ουκρανία, αλλά η Ρωσία απέτυχε η Ουκρανία, η κυβέρνηση Ουκρανίας είναι ακόμα στην εξουσία. Και Βεβαίω η βασική ανησυχία του Κρεμλίνου όσον αφορά την βιωσιμότητά του, δηλαδή δίπλα σε μια δημοκρατική Ουκρανία, έχει πλέον ε, επιβεβαιωθεί. Σε αντίθεση με τις αποτυχίες στην Ουκρανία, η παρέμβασή της στην Συρία ήταν επιτυχία σύμφωνα με τα δικά της ε, μέτρα. Επέδειξε μια τακτική χρήση ισχύω ε, εδραίωσε τη θέση της ως μεγάλη δύναμη, σταθεροποίησε το καθεστώς Άσαντ ε, και βεβαίως υπήρχαν και μεγάλες μάζες προσφύγων που έφευγαν από την βαρβαρότητα του Ασάντ. Συνεχίζονται λοιπόν οι πολιτικέ ε, ε, που ακολουθεί η Γεωργία και στην ε, Ουκρανία. Εκεί πέρα προσπάθησε να μην υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ μέσω της χρυσή βία και αποσχιστικών κίνηματων. Η Στρατηγική Εθνική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015 κατηγορεί ρητός την επέκταση του ΝΑΤΟ ω ασφάλεια, ως απειλή για τη ρωσική ασφάλεια. Και ζητάει ακριβώ να ακολουθηθούν ή παραδοσιακές μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί η εξωτερική ιδεολογία. Και τώρα οι Ρώσοι θύνοντες θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Άτο τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και ζητούν ακριβώς μια να καταστήσουν τα θεσμικά μας όργανα ένα κενό κέλφος και όμως αντιμετωπίζουν ένα ΑΕΠ περίπου ανάλογο με αυτό της ε, Νότιας Κορέας με ανεμική ανάπτυξη και δεν μπορούν να προσελκύσουν ακόλουθους ε, στο μοντέλο τους. Εξακολουθούν να έχουν μια ικανή στρατιωτική μηχανή που τους δίνει την δυνατότητα να διαταράσουν αυτήν την φιλελεύθερη διεθνή τάξη, αλλά δεν μπορούν να την ανατρέψουν. αυτού η Ρωσία θα συνεχίσει ευκαιριακά να εκμεταλλεύεται στρατηγικέ ευκαιρίε ε, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, στο Αφγανιστάν για να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη και την Δύση. Η παραμονή του Προέδρου Πούτιν ε, μετά τις εκλογές ε, του Μαρτίου 2018 μας λέει πως οι πολιτικές αυτές θα συνεχιστούν μεσοπρόθεσμα και θα απαιτήσουν μια απέντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τελειώσω με λίγα λόγια για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής. Βεβαίως, ε, όπως ανέφερε και η Μαρία, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε πέντε αρχές ε, που μπορούμε να περιγράψουμε ως ένα μείγμα αυστηρότητας και επαφών και μπορούμε να πούμε το εξής, να τους αντιμετωπίσουμε όπου πρέπει και να συνεργαζόμαστε και όπου μπορούμε. έχουμε ένα μείγμα λοιπόν συνεργασίας και αντιπαλότητας ε, και παραμένει σωστή αυτή η προσέγγιση. Επίσης θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την στενή συνεργασία με τους εταίρους στο G7. Αυτό έχει λειτουργήσει ήδη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το ότι υπάρχουν οι προσπάθειες ε, της Ρωσίας για να διχάσουν την Ευρώπη και την Ατλαντική κοινότητα, οι οποίες έχουν αποτύχει και έχουν οδηγήσει σε συσπήρωση της ε, Δύσης αλλά αυτό δεν συνέβη αυτομάτως και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Πρέπει ε, αντιθέτως να συντονιζόμαστε συνεχώς. Μέσω πρόθεσμα οι ευρωπαϊκές σχέσεις με την Ρωσία θα παραμένουν περιορισμένες σε κάποια κέρια συμφέροντα όπως η αντιτρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή και η μη διάδοση πυρηνικών. Τελικά οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής Ρωσίας, δηλαδή να προστατευθεί το καθεστώς που από εσωτερική αντιπολίτευση και να δρά ως μεγάλη δύναμη και η Ρωσία θα πρέπει να αλλάξει την επιθετική της ε, φύση, αλλά αυτό δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί, καθώς αυτός ε, ο στόχος πηγαίνει ενάντια στους ε, στόχους του Κρεμλίνου για να παραμείνει στην εξουσία ως αυταρχικό Αλλά αυτόν τον στόχο πρέπει να ακολουθήσουμε, καθώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει αποφασιστική και η προσπάθεια αυτή σημαίνει ότι θα γίνεται άργα και σταθερά. Και βεβαίως ε, αυτό είναι μειονέκτημα και πλεονέκτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί να σχηματίσει κάποια πολιτική, αλλά όταν το κάνει την ακολουθεί σταθερά. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις παρατηρήσεις. Έχουμε εξαντληθεί από ό,τι φαίνεται, λέει ο πρόεδρος. Σάντρα, εσείς πρώτοι. Να ακούσουμε και τα συμπεράσματα σας. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Η κυρία Καρνιέτε. Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι μπορούν να αντιληφθούν την πολιτική της Ρωσίας, άλλοι από το εσωτερικό, άλλοι από το εξωτερικό και σε αυτούς έχει βασιστεί η έκθεση. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι είναι δύσκολο να προετοιμάσει κανείς μια έκθεση για τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας σε αυτό το στάδιο, όπου ουσιαστικά έχουμε μια πολιτική σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη πόλεμος. Γιατί δεν μου αρέσει να τη χρησιμώ ελαφρά την καρδία. Γιατί χρησιμοποιείται για κάτι πολύ σοβαρό, για την άμυνα των χωρών μας. Αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ σε πολύ σοβαρά δημοσιεύματα. Όταν έχουμε έναν Υπουργό Άμυνας χώρας του ΝΑΤΟ, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός κυβερνοπολέμου με τη Ρωσία και, και μιλώ για τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας. Ορισμένοι μπορεί να είπαν ότι υπερέβαλε, αλλά στην πραγματικότητα παρουσιάζει πραγματικά την κατάσταση της σχέσης μας με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκρούσεις και ανταγωνισμό αναφερόταν στις, ε, ε, στις κυβερνοεπιθέσεις ε, από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στην υπηρεσία για τα χημικά όπλα στη Χάγη. Και είχαμε και παλαιότερες τέτοιες, τέτοια περιστατικά, hacking από ρωσικές υπηρεσίες στο σύστημα GPS κατά τη διάρκεια στρατιωτικών κινήσεων στη Φινλανδία. Ας μην έχουμε, ας μην είμαστε Έχουμε μπροστά μας μια σύγκρουση στην οποία χρησιμοποιούνται και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα με τρόπο ενοποιημένο προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι. Αυτή είναι, αυτός είναι ο κίνδυνος. Η Ρωσία δεν είναι η μόνη που χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία. Τα χρησιμοποιούν και άλλα ε, αυταρχικά, πολιταρχικά καθεστώτα και εδώ έρχεται η συζήτηση την οποία ορθά επεσήμανε ο εκπρόσωπος, ο υπηρογνώμονάς μας ε, για το ζήτημα της χρήσης αυτών των εργαλείων από απολυταρχικά καθεστώτα και έρχεται και η συζήτηση για το τι συμφέρει στο Ιράν, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε αυτές τις επιθέσεις, αλλά επίσης θα πρέπει να προετοιμαστούμε να αναλάβουμε και δική μας δράση εκ των προτέρων, προκειμένου να ε, αποθαρρύνουμε την πιθανότητα τέτοιων επιθέσεων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε έναν κοινό ορισμό για αυτό τη νέα μορφή σύγκρουση στην οποία εμπλεκόμαστε. Δεν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες ή κανόνες που να ρυθμίζουν τον κυβερνοχώρο, ούτε τη συμπεριφορά σε αυτόν. Και υπάρχουν και άλλες πτυχές της σύγκρουσης με την ε, Ρωσία. Έχουμε πράκτορες από τη Ρωσία, από τις μυστικές τους υπηρεσίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Σέλισμπρου, είδαμε να ενεργούν. Δεν πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο να πρωταγωνιστούν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι μια σύγκρουση στην οποία ουσιαστικά πρωταγωνιστούν οι μυστικές υπηρεσίες και το περιβάλλον του Προέδρου της Ρωσίας. Ε, αξιοποιούνται επικοινωνιολόγοι, ε, ε, αξιοποιούνται οι φόβοι, οι ψευδείς ειδήσει, ψευδείς, ισχυρισμοί που έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικοί από τα τάγκς. Χρειάζεται μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα ρωσική απειλή, αυτή την ρωσική κούκλα με τις πολυεπίπεδες απειλές την οποία περιέγραψε και, περιέγραψαν και οι δύο εμπειρογνώμονες μας. Όμως, ταυτόχρονα έχουμε επίσημους αναλυτές όπως ο Καραγκάνοφ οι οποίοι ξεκάθαρα μιλούν ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει και θερμή πολεμική σύγκρουση, η οποία, ο οποίο αναφέρει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να προετοιμαστεί για την πιθανότητα ενός πραγματικού πολέμου και ότι θα πρέπει η Ρωσία να συνεργαστεί και να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση ω εταίρο τη για, τα θέματα τη ασφάλεια για να προλάβει ένα τέτοιο πόλεμο. Έρχεται εδώ λοιπόν και η συζήτηση για αυτήν την πολύ σοβαρή συζήτηση για την δημιουργία ενό ευρωπαϊκού στρατού. Αυτή η ιδέα προσλαμβάνεται πολύ διαφορετικά στη Μόσχα από ότι στην Ουάσιγκτον. Στην Ουάσιγκτον το θεωρούν τον Ευρωπαϊκό στρατό ως έναν τρόπο να υποβαθμιστεί το ΝΑΤΟ. Και επιθυμούν ενίσχυση του, του ρόλου του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας, ενώ στη Ρωσία ε, γίνεται καλο, είναι καλοδεχούμενη αυτή η ιδέα του Ευρωπαϊκού στρατού. Έρχομαι τώρα στο ποιε πρέπει να είναι οι πολιτικέ μα. Έχουμε υιοθετήσει, όπω αναφέρθηκε, τι πέντε αρχέ το 2016 για την πολιτική μα έναντι τη Ρωσία. Θα πρέπει αυτέ οι αρχέ να μεταφραστούν στην πράξη και να έχουμε περισσότερες σχέσεις σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με την ε, Ρωσία. Δεν θέλω όμω να χρησιμοποιήσω το λόγο συνεργασία ούτε, τον όρο διάλογος. Γιατί για να μιλήσει κανείς για συνεργασία και διάλογο πρέπει να έχει δύο μέρη που και τα δύο να το επιθυμούν. Νομίζω ότι το πιο ακριβή ε, ορολογία θα ήταν να μιλήσουμε για διαβουλεύσεις και για επικοινωνίες. Η επιλεκτική ε, συζήτηση με τους Ρώσους θα έχει περισσότερο ως στόχο την διαχείριση του status quo και να απομακρύνουμε την πιθανότητα της κατάρρευσής του ή της διάβρωσης του. Έχουν αναφερθεί διάφοροι τομείς στους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε με τους Ρώσους έχουν προκύψει εν μέρη από το δίκτυο ε, των ειδικών για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Για παράδειγμα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ε, που είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή του Ντόμπασκ, ε, για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή αυτή. Επίσης, έναν υψηλού επίπεδου διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή και Ρωσίας για την Κεντρική Ασία. Η αξιοποίηση των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και συμφωνιών σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Ασία, την Κίνα επίση. και το πώς να αξιοποιήσουμε τον λεγόμενο νέο δρόμο του μεταξιού. Ένα άλλο θέμα μπορεί να είναι η συνεργασία μας για την αντιμετώπιση του νέου προγράμματος για τα πυρηνικά του Ιράν. Ε, εδώ είναι ένα τομέας στον οποίο συμφωνούμε με την Ρωσία. Συρία υπάρχουν ε, αντιφατικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, βρούμε από κοινού το δρόμο για την ε, ειρήνη. Υπάρχουν επίσης παιδεία όπως είναι η η κλιματική αλλαγή, αρκτικός κύκλος, θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ε, πρόκειται για θέματα τα οποία δεν έχουν επηρεάσει, ας πούμε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω ε, του, της του παγώματος των σχέσεων κλπ. Ε, επίσης ε, το θέμα της των επαφών με την ε, κοινωνία των πολιτών, με τους πολίτες, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Ε, η Μαρία Μενδράς αναφέρθηκε επίσης ε, και σε θέματα διαλόγου επί αμφιλεγωμένων θεμάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε σωστά μέτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους μας που εξέφρασαν την άποψή τους όσον αφορά αφορά το θέμα αυτό και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί από κοινού θα μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε, να εκπονήσουμε μια καλή ε, έκθεση η οποία θα είναι σε θέση να που θα είναι ικανή να παρουσιάσει τα πραγματικά προβλήματα αλλά και τις ελπίδες μας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, Σάντρα Καλνιέτε, θέλετε εσείς να απαντήσετε. Ίσως να πω δύο λόγια, λέει ο το 2015 το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο είναι αρκετά καλό, είναι πραγματικά καλό και το απέδειξε αυτό τα τρία τελευταία χρόνια. Εγώ δεν θα άλλαζα υπερβολικά το γενικό πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ήδη οικοδομηθεί. το 2014 και το 2015 όταν ασχοληθήκαμε, αντιμετωπίσαμε το θέμα, ίσως ε, είχαμε και περισσότερες ελπίδες ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν πορεία ή να βελτιωθούν. Ε, εδώ όμως ε, βλέπουμε ότι τα προβλήματα επιμένουν και ίσως στο νέο ψήφισμα θα πρέπει αυτό να φαίνεται. Επίσης, η G 7 και η Διαθενική Συμμαχία για την ε, Ρωσία δίνουν κάποια στοιχεία όσον αφορά την ε, πολιτική, γιατί μεμονωμένα ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να επιτύχει, αλλά συλλογικά ναι, μπορεί κάτι να γίνει. Τέλος. Η στρατηγική για τη Ρωσία θα δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Είτε πρόκειται για την ενωσιακή, είτε πρόκειται για την διατλαντική ε, στρατηγική. Επομένως, εάν ε, αναφέρεστε σε συγκεκριμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, του κράτους δικαίου, επίσης παροχή συμβουλών σχετικά με την θεσμική δημοκρατική εξέλιξη της ε, Ρωσίας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ψηφίδες ε, της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε, που συμμετείχατε σε αυτήν την ε, συζήτηση. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση, αλλά έχουμε άλλα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ε, στις 26 ε, Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου θα, γίνει, θα γίνουν οι επόμενες συνεδριάσεις. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Βγείτε έξω, χαρείτε τον ήλιο, να περάσετε καλά και τέλος της συνεδρίασης.